to the afternoon Συνεχίζουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ψηφίσουμε σε λίγο, αλλά στο μεταξύ καθίστε. Με γρήγορα παρακαλώ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη σήμερα το απόγευμα. Πρώτα θα ψηφίσουμε το σχέδιο κειμένου ε, για τον προπολογισμό Πατέρα και Γιάρ. Συγγνώμη, θέματα, ε, θέματα προστασίας των παιδιών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια των εργασιών μας διαπιστώσαμε ότι η κινητικότητα των πολιτών έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα και πολλές ε, διανέξεις σε σχέση με τα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν είναι, που έχουν έρθει εδώ και τα έχουμε δει, μας προβλημάτισαν πολύ. Υπάρχει λοιπόν ε, η πρόταση για ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την προστασία των παιδιών που προτείνει η Επιτροπή μας. Η Επιτροπή λέει ότι το δικό μας ε, πιλωτικό σχέδιο καλύπτει το θέμα της δικαιοσύνης και επικαλύπτεται με άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις οικογένειες. Εδώ όμως πρέπει να τονίσουμε ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι πιστική. Έχουμε κοιτάξει, τι λέει το πόρταλ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δικαιοσύνη, αναφέρει τα θέματα των διαζυγίων, ε, το θέμα της διατροφής, και το θέμα των παιδιών και πώς θα γίνεται σεβαστή επιθυμία των παιδιών. Έχουμε λοιπόν την αίσθηση ότι το δικό μας το σχέδιο δεν επαναλαμβάνει τις πληροφορίες που υπάρχουν στο πόρταλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα για την προστασία των παιδιών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να ασχοληθούμε εμείς περισσότερο και έχουμε την αίσθηση ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι μηχανισμοί στήριξης είναι στη διάθεση των γονιών. Πάντα για την προστασία των παιδιών. Υπήρξε μια ερευνητική αποστολή στη Δανία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία για αυτό το θέμα και δημιουργήθηκε και μια ομάδα εργασίας και είχαμε και ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω λοιπόν ότι αν συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν ε, στη, στο πόρταλ της δικαιοσύνης, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε. Δεν επαναλαμβάνουμε πληροφορίες που ήδη υπάρχουν, επαναλαμβάνω. Προσθέτουμε επιπλέον ε, πληροφορίες αυτές που υπάρχουν στο πόρταλ. Είτε τις συμπληρώνουμε αυτές που ήδη υπάρχουν, είτε προσθέτουμε άλλες. Ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διχάζονται απόψεις και όταν ετοιμάσαμε το σχέδιο αυτό ήρθαμε σε επαφή με τον κόσμο που είναι υπεύθυνοι για τις υποθέσεις των παιδιών και οι αξιωματούχοι τα ξέρουν και συμφωνούν μαζί μας ότι λείπουν πληροφορίες που σχετίζονται με τις αναφορές αυτές που παίρνουμε. Η μονάδα δικαιοσύνης πάντως τελικά θα αποφασίσει αν θα μπει στην κατηγορία Γ ή όχι. Εμείς δεν συμφωνούμε με τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες πρέπει να είναι, που είναι τώρα στο πόρταλ της δικαιοσύνης, πρέπει να συμπληρωθούν από αυτά που έχουμε εμείς να προσθέσουμε. Γι' αυτό και ζητάω τη στήριξη των συναδέρφων στην προσπάθεια αυτή να την υπερψηφίσουν. Είναι ένα σχέδιο που θα συμπληρώσει τη δουλειά που ήδη εκπονεί η Επιτροπή μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πιτέρα. Τώρα, συνεχίσουμε. περνάμε στην ψηφοφορία. Υπέρ, παρακαλώ. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Ηλεκτρονικά για να έχουμε ακριβώς τα νούμερα. Ψηφίστε, παρακαλώ. Ε, από το ΕΛΚ ψηφίζουν παραπάνω από όσοι μπορούν. Ένας παραπάνω, εντάξει, ένας παραπάνω τώρα είναι μόνο. Ωραία, τώρα είναι εντάξει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε με ομοφωνία. Συγχαρητήρια. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, Τώρα που το εγκρίναμε αυτό εδώ στην Επιτροπή μας, θα υποβληθεί ως τροπολογία από την Επιτροπή μας στην Επιτροπή Προεπολογισμών, η οποία θα το ψηφίσει αργότερα. Μην ξεχάσετε τις κάρτες, τα μηχανήματά σας, έτσι. Και συνεχίζουμε. Όπως θα θυμόσαστε πριν από τη μεσημεριανή διακοπή, Είχαμε κάποια πρακτικά ζητήματα σχετικά με το σημείο 17, αναφορά 1053 σχετικά με έργο κατασκευής δεξαμενής ρύθμισης για τον ποταμό Σεβέζο. Δεν μπορούσε να είναι εδώ έγκαιρα η αναφέρουσα, αλλά τώρα είναι εδώ. Οπότε θα δώσω το λόγο στην Κιάρα Ποσέλη για πέντε λεπτά το πολύ. Παρακαλώ. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ανάφορων Καλημέρα, λέγομαι κ. Μποζέλη και είμαι αναφέρουσα της ε, αναφοράς 153-2016 ε, από την περιοχή Παπατζοβάνη του Μπρέσο. Όπως θα δείτε στο φιλμ ε, που βλέπετε στην οθόνη, τέσσερα εκτάρια του Βόρειου Πάρκου θα καταστραφούν και θα τοποθετηθεί τσιμέντο για να δημιουργηθεί ένα χώρο βάθους 10 μέτρων όπου χωράει 38.000 τετραγωνικά μέτρα ε, και δεν μπορεί να δεχτεί 250.000 κυβικά μέτρα νερό βρόχινο μόλις 30 ε, μέτρα από την γειτονιά μας την ε, πυκνοκατοικημένη Παπατζοβάνη όπου υπάρχουν διάφορα σχολεία και παιδικές χαρές ο κίνδυνος είναι μεγάλος, διότι στις 28 Ιουνίου η Περιφέρεια της Λαμβαρδίας κατά τη διάσκεψη των υπηρεσιών ενέκρινε το τελικό σχέδιο της δεξαμένης ρύθμισης. Παρ' όλα αυτά ε, κρεμούν δύο αποφάσεις του δικαστηρίου ε, από τη Ρώμη ε, που έχουν υποβληθεί από το Δήμο του Μπρέσο. Η βιοπικιλότητα αυτού του πάρκου είναι ευρεία. Στο βίντεο και στις φωτογραφίες μπορείτε να παρατηρήσετε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία θάμνων και δέντρων και φυτών στο πάρκο για να μην μιλήσουμε για την Πανίδα έχουμε πολλά ε, πτηνά, ε, χίνες, ε, πάπιες, διάφορα είδη πτηνών, παπαγάλους, λαγούς και πολλές πεταλούδες. Στο το πάρκο επισκέπτονται καθημερινά οι περιοίκοι και πριν από λίγα χρόνια τοποθετήθηκε και μια γέφυρα που συνδέει αυτά τα 4 εκτάρια πάρκου με το ευρύτερο πάρκο στην περιοχή Μπρουτσάνο, στη βόρεια πλευρά της, ε, του Δήμου του Μιλάνου. Οι βασικοί λόγοι που αντιτιθέμεθα στην κατασκευή της δεξαμένης είναι διάφοροι. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να διαφυλάξουμε το πάρκο μας ε, που αποτελεί πηγή οξυγόνου, το Βόρειο Πάρκο μεταξύ άλλων. Το 2017 έλαβε από το Συμβουλίο της Ευρώπης ε, τον ειδικό χαρακτηρισμό ε, τοπίου και ε, δύο εκατομμύρια επισκέπτες έχει κάθε χρόνο και θεωρούμε ότι πρέπει να το προστατεύσουμε. Γι' αυτό έχουμε συλλέξει περίπου 3.000 υπογραφές πολιτών που αντιτίθενται στην καταστροφή αυτού του πάρκου και που υποστηρίζουν τη μάχη μας. Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι τα ύδατα που θα συλλέγονται για πολλές μέρες στην δεξαμενή θα προέρχονται από ένα πολύ μολυσμένο ποτάμι που περιέχει επικίνδυνες ουσίες όπως το γλυφοζάτ που έχει απαγορευτεί σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως για παράδειγμα στη Γαλλία και που υπάρχει στο Σεβέζο με τον μεταβολίτη του ε, σε περιεκτικότητα 100 φορές πάνω από την οριακή τιμή. Υπάρχουν και άλλες επικίνδυνες ουσίες όπως ε, το εξασθενές χρώμιο το οποίο έχει καταταχθεί ως ε, ε, καρκινογενές. Η τοξική ύλη ε, που θα αποτίθεται θα δημιουργήσουν προβλήματα στον αέρα και θα είναι τεράστιο το κόστος για τη διάλυση αυτών των τοξικών λιμάτων που μπορεί να μείνουν εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα με επιβλαβή συνέπειες για την υγεία όλων μας. Εάν συνεχιστεί εάν καθαρίζαμε το ποτάμι θα ήταν λιγότεροι κίνδυνοι τα 1400, ε, αν καθαρίζαμε τους 1.400 χώρους ε, απόθεση απορριμμάτων που υπάρχουν κατά μήκος του ποταμού ε, θα μπορούσαμε να εκτρέψουμε το ποτάμι προς άλλη κατεύθυνση αλλά αυτό δεν γίνεται, το ποτάμι αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά μολυσμένο και ο Δήμος αντιτίθεται σε αυτό Επίσης προβλέπεται, προβλεπόταν αρχικά η κατασκευή πέντε δεξαμενών για τα ε, παραπάνω ύδατα του ποταμού. Ε, αυτό το ο Βόρειο Πάρκο ήταν η τελευταία λύση που είχε προβλεφθεί και που είχε τη χαμηλότερη χωρητικότητα. Μόνο δηλαδή το 5% του συνολικού όγκου. Διάφορε γνωμοδοτήσεις ειδικευμένων τεχνικών υποστηρίζουν επίσης ότι το σύστημα των δεξαμενών ούτω ή άλλω δεν θα αρκούσε για να αντιμετωπιστούν οι πλημμύρε, αφού και γι' αυτό το έργο έχει αλλάξει ε, τόσο χρονικά όσο και χωρικά. Η κατασκευή των δύο μεγαλύτερων δεξαμενών που θα υποδέχονταν το μεγαλύτερο ποσοστό, ποσό των υδάτων ε, έχει αναβληθεί λόγω ε, μιας μολυσμένης περιοχής που πρέπει να καθαριστεί. Ε, και έτσι το έργο έχει καθυστερήσει σημαντικά. Επίσης η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών ε, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα επέλυε το πρόβλημα, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Επίσης, εμείς ε, οι κάτοικοι της περιοχής έχουμε υποστεί οικονομική ζημία, διότι οι αξίες των κατοικιών μας έχουν μειωθεί σημαντικά. Επίσης για την κατασκευή της δεξαμενής, η οποία θα διαρκέσει περίπου τρία χρόνια, φαντάζεστε πόσο προβλήματα θα δημιουργήσει στην περιοχή μας, διότι θα αυξηθεί η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, η παρουσία σκόνης και θα αυξηθούν και οι κραδασμοί. Οπότε θέλουμε την υποστήριξή σας ε, για να αντιταχθούμε σε αυτό το σχέδιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρου όλων των πολιτών της περιοχής μου, τα μέλη της Επιτροπής αυτή και ειδικότερα τον κύριο Αλμπέρτο Τσίριο και το προσωπικό του που έδωσαν σε απλούς πολίτες της Ευρώπης τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την επιχειρηματολογία τους κατά ε, της δεξαμενής αυτής ε, ε, ρύθμισης ε, για τον ποταμό Σέβεζο και ευχαριστώ και τους συνεργάτες που μου έδωσαν τη δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για αυτές τις ε, πληροφορίες. Ε, Στρέφουμε στην ε, Επιτροπή, κυρία Προύνα, να μας δώσει περαιτέρω εξηγήσει σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα. Αυτά τα υδραυλικά έργα τα οποία προτίθενται για την αποθήκευση λιγότερων από 10 δισεκατομμυρίων γαλονιών νερού, όπως δηλαδή εδώ και στην προκείμενη περίπτωση, εμπίπτουν στο παράτημα 2 της οδηγίας EIA. Και αυτό σημαίνει ότι αυτού του είδους τα, τα project ε, πρωτού εγκριθούν ε, μπήκουν στην διαδικασία ε, εποπτείας της, που προβλέπεται στην οδηγία EIA με βάση το άρθρο 4. Ο ο στόχος αυτής της παρακολούθησης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο το εν λόγω έργο ε, δύναται να έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και κατά συνέπεια αν ε, χρειάζεται μια πλήρης διαδικασία εξέτασης ε, στο πλαίσιο του EIA ή όχι. Άρα λοιπόν έπεται ότι η έγκριση αυτής της, αυτών των έργων για τη μείωση των υδραυλικών έργων για τον ε, ποταμό Σεβέζο, χωρί να υπάρχει πλήρη ERA, δεν ε, συνιστά παραβίαση τη ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσία. Οι πληροφορίε από την αναφέρουσα δεν περιλαμβάνουν κάποια στοιχεία τα οποία να επιτρέπουν στην Επιτροπή να ε, τεχμέρει ότι η εξέταση μέχρι στιγμή δεν έχει λάβει χώρα για το εν λόγω έργο ή ότι δεν προτίθεται οι αρμόδιε εθνικέ αρχέ να προβούν σε μια τέτοια εξέταση μελλοντικά, προτού δηλαδή εγκρίνουν το έργο. Θα πρέπει επίση να ληφθεί υπόψη ότι στο πλαίσιο των λόγων διαδικασιών οι αρμόδιες εθνικέ αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλα τα σχετικά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στο, άρθρο, στο παράδειγμα 3 τη οδηγία, μεταξύ άλλων τις, ε, τα χαρακτηριστικά των έργων, δηλαδή δυνητικές επιπτώσεις ε, στην ε, μορφολογία του εδάφους, στην κλωρίδα και πανίδα, τον κίνδυνο ατυχημάτων και ούτω καθεξής. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι τέτοιου είδους έργα που είναι απαραίτητα δηλαδή για την αποκατάσταση υποτιθέμενων μολυσμένων εδάτων μπήκτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Το οι αρμόδιες λοιπόν εθνικές ε, ε, μυστικές και δικαστικές αρχές είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του σχετικού άρθρου ε, της οδηγίας και θα πρέπει να αναλαμβάνουν την αποκατάσταση περιπτώσεων όπου ακριβώς υπάρχει τέτοιου είδους παραβίαση της νομοθεσίας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, ο λόγος τώρα στους συναδέλφους, αλλά κυρία Σέβη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την αναφέρουσα για αυτή την αναφορά που παρουσίασε. Να την ευχαριστήσω για όλες τις υπογραφές που συνέλεξε προς υποστήριξη αυτού του έργου που είναι το χιλιοστό που βλέπουμε να αντιτίθεται στα προβλήματα που πάνε να δημιουργηθούν σε μια περιοχή στην επαρχία του Μιλάνου που εγώ γνωρίζω καλά διότι και εγώ ζω εκεί κοντά. Το χιλιοστό λοιπόν έργο που προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα ε, αυτό της τσιμεντοποίησης παντού με, άλλ, με τσιμέντο άλλου είδους ε, ουσιαστικά με την κατασκευή δεξαμενών ρύθμισης αντί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα το υδρολογικό που πλήττει την περιοχή εκείνη με άλλο τρόπο διότι είναι σαφές ότι ο ποταμός ε, Σέβεζο κατά διαστήματα συμπεριφέρεται περίεργα διότι οι βροχές ε, και τα νερά δεν απορροφώνται παρκώς από τα εδάφη με σωστό τρόπο. Αυτό γιατί λόγω της ε, τεράστιας χρήσης τσιμέντου που έχει γίνει άναρχα τις τελευταίες δεκαετίες. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια λύση κατασκευάζοντας αυτές τις δεξαμενές που από όσο καταλάβα εγώ από την παρουσίαση της αναφέρουσας. Οι δεξαμενές αυτές ε, είναι λάθος προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος ε, και σίγουρα μη βιώσιμες, ε, δημιουργώντας διάφορα προβλήματα τα οποία θα επιβαρύνουν την κατάσταση. Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι όλα αυτά εξαρτώνται από το κράτος μέλος και από αυτό εξαρτάται να γίνουν σωστά τα πράγματα, εγώ θα ήθελα να απαντήσω στην Κομισιόν ό,τι αναφέρωσα. Δεν έθεσε το θέμα μόνο το περιβαλλοντικό, αλλά και την πιθανή μόλυνση των υδάτων μέσα σε αυτές τις δεξαμενές. Γι' αυτό δεν έχουμε κανένα στοιχείο στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγγνώμη. Και όπως φαίνεται οι εθνικές αρχές και οι τοπικές αρχές ε, τα βλέπουν όλα ρόδινα. Ωστόσο δεν έχει έτσι. Στην εκτίμηση αντικτύπου που έγινε για το έργο ε, λένε ότι η ποιότητα των υδάτων έχει χαρακτηριστεί ως άσχημη. Ε, όχι μόνο περιέχει, όπως είπε αναφέρουσα, γλυφόσατ σε ποσότητες επικίνδυνες, αλλά και βαρέα μέταλλα, όπως εξασθενές χρώμιο. Όλα αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, όλες αυτές οι ουσίες που είναι τοξικές και επιβλαβείς, θα συνεχίσουν να υπάρχουν σε αυτά τα υδατά, σε αυτές τις δεξαμενές ρύθμισης και μπορεί να ε, ε, βρεθούν και στην ατμόσφαιρα όταν θα αποξηραίνονται αυτές οι δεξαμενές. Οπότε εμείς στραφήκαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε κατά πόσο τα νερά αυτά, τα λιμνάζοντα θα επηρεάζουν την υγεία και μας είπαν δεν έχουμε στοιχεία διότι τα κράτη-μέλη, η Ιταλία στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα δεν έχουν υποβάλει τα σχέδια διαχείριση των δεξαμενών ρύθμιση ε, και των λεκανών απορροή. Ε, τελικά έχουμε αυτά τα στοιχεία. Πείτε μα, Κομισιόν, ε, πότε θα μπορέσουμε να τα έχουμε, διότι βρισκόμαστε, όπω είπα, στο χιλιοστό έργο που θα καταπατήσει τα δικαιώματα των ανθρώπων και την υγεία του. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Πρόεδρο να διατηρήσει ανοιχτή την αναφορά και επίσης να ζητήσω να γίνει και μια μελέτη στην Ευρώπη για το πώς το πρόβλημα αυτό της παρεκτροπής των ποταμών ε, ε, των υδάτων των ποταμών ε, πώς έχει λυθεί όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και αλλού στην Ευρώπη στο να βρούμε ποιες είναι οι βελτιστές πρακτικές που κατά την άποψή μου θα υπάρχουν σε σχέση με αυτά τα τρελά έργα που προτείνεται εδώ ε, και τα οποία δεν έχουν κανένα οικονομικό συμφέρον και είναι απολύτω αναχρονιστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σπουλιέζα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να χαιρετήσω και εγώ εκ μέρους του κυρίου Αλμπέρτο Τσίρι, ο οποίος ζητά συγγνώμη για την απουσία του, αλλά έγινε άθελά του. Είχε προγραμματίσει ήδη την πτήση του στις 3.40. Άκουσα πολύ προσεκτικά την αναφέρουσα και συμφωνώ με τα όσα μας είπε. Κάτι που στηρίζεται και από τις εικόνες που είδαμε. Εδώ σίγουρα δεν είναι, δεν το σωστό σημείο για να τοποθετηθούν δεξαμενέ ρύθμιση. Θα είναι τεράστια υπεραβολητική ζημιά και θα υπάρξουν και δομικά προβλήματα στα κτίρια που βρίσκονται κοντά. Ε, φυσικά θα πρέπει να γίνει η γνωμοδότηση του κ. Τσίριο ε, που να προτείνει λύσεις λιγότερο προβληματικές. Ε, έχουμε και πολλές επιφυλάξεις ε, όσον αφορά τις ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιφέρεια της Λομβαρδίας. Λέμε λοιπόν να στείλουμε μια επιστολή στην Λομβαρδία, στην περιφέρεια, για να τους πούμε να επεξετάσουν τις εναλλακτικές, να δουν αν υπάρχουν άλλες τεχνικές λύσεις με τις οποίες θα συμφωνεί και ο πληθυσμό. Ζητώ και εγώ η αναφορά να μην είναι ανοιχτή, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε το... την υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Uh... Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, συμφωνώ με τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Απλώς θα ήθελα να ε, υπογραμμίσω κάτι που ανέφερε η Επιτροπή. Μια πρόταση, η οποία θεωρώ πως είναι ζωτική σημασία. Είπε λοιπόν η Επιτροπή ότι δεν μπορεί κανείς να συμπεράνει αυτόματα κάτι. Ναι, ε, προφανώ εντάξει. Αλλά αν δεν έχουμε λοιπόν αρκετό χρόνο για να το κάνουμε αυτόματα, τότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε αυτό το χρόνο. Θα πρέπει δηλαδή να διερευνήσουμε ε, επί τούτου τι ακριβώς συμβαίνει. Σε διαφορετική περίπτωση ε, απλώς θα βρεθούμε στη θέση του να πούμε ότι παθητικά αποδεχόμαστε τα πράγματα όπως έχουν και δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν μία γνωμοδότηση από τη δική μας ε, πλευρά, είτε αρνητικά είτε θετικά εννοούμενη, οπότε θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά προκειμένου ακριβώς να διευκρινιστεί αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Άρα λοιπόν ολοκληρώσαμε με τους ομιλητές και δίνω και πάλι το λόγο στην αναφέρουσα, την κυρία Μποσέλη, για δύο ακόμα λεπτά κατά το μέγιστο. Ε, Πολύ απλά ήθελα να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν και άλλα έργα χαμηλότερου κόστου, πιο καινοτόμα, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι δεξαμενέ ρυθμίσεις, πέραν του ότι κοστίζουν πολύ οικονομικά, είναι κατασκευέ απερχαιωμένε. Διότι ξέρουμε ότι πέραν των υδραυλικών προβλημάτων Ε, που παρουσιάζουν υπάρχουν άλλες ε, λύσεις για το πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε τις απόψεις κάποιων εμπειρογνωμόνων ε, επί του θέματος που ενδεχομένως θα μπορούσαν να ρίξουν μια ματιά πάλι στο έργο για να δουν αν υπάρχει ένας άλλος τρόπος επίλυσης του προβλήματο με τις πλημμύρες στον ποταμό Σέβεζο. Και σίγουρα θα μπορούσαν να μας προτείνουν κάτι άλλο ως λύση. Αυτό, διότι εδώ το έργο αυτό θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, καταστρέφει 4 εκτάρια πάρκου. Ευχαριστώ. Thank you very much. And... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Για να ζητήσω την άψη της Κομισιόν με μεγαλύτερη ακρίβεια η εξολόγησή σας είναι επί της διαδικασίας ή επί της ποιότητας του έργου. Μπορείτε να με εξηγήσετε εσείς διαδικαστικά το εξετάζετε ή έχετε μπει και έχετε εξετάσει και ε, το έργο και επί της ουσίας είναι αρμοδιότητα δική σας αυτό ήθελα να μάθω διότι πραγματικά ναι συνήθως εστιαζόμαστε μόνο στις διαδικαστικές πτυχές αλλά φυσικά αν έχουμε σαφή αποδεικτικά στοιχεία παράβασης ε, το αφορούν της ποιοτικές πτυχές ε, της εξολόγησης φυσικά μπορούμε να εξετάσουμε και αυτές Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε διάλογο μεταξύ των δυο σας αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό τώρα, θα διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να στραφώ στην αναφέρουσα και να πω ότι δεν τελειώνουν εδώ τα πράγματα, δεν έχουν καν αρχίσει. Ε, μόλις αρχίζουν μάλλον. Ε, θα στείλουμε μια επιστολή στην περιφέρεια Και το επόμενο βήμα είναι ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε τους συντονιστές, δηλαδή τους ηγέτες των διαφόρων ε, τους εργούς των διαφορών ομάδων στην Επιτροπή για να δούμε αν μπορούμε να αναθέσουμε, να γίνει μια μελέτη ε, για να δούμε πώς θα μπορούσε να επιληθεί αυτό το πρόβλημα των πλημμυρών, άλλες βέλτιστες πρακτικές που έχουν ε, εφαρμοστεί στο παρελθόν αλλού, να κάνουμε έναν απολογισμό του πού, βρισκόμαστε, να οργανώσουμε κάποια ακρόαση, ή να αναθέσουμε κάποια άλλη μελέτη μες στις επόμενες ημέρες. Οπότε θα το συζητήσουμε μεταξύ συντονιστών και φυσικά αν θέλετε μπορούμε να στείλουμε μια, επιτροπή, μια επιστολή ενημερωτική στην Επιτροπή Ένβη. Ε, ε, Βλέποντα την Ελεονόρα να σηκώνει το χέρι τη, ξέρω τι θέλετε να Δεν χρειάζεται να πάρετε τον λόγο. Το είπα. Αυτό να κάνουμε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Εύε. Ναι, ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να μάθω. Είπατε θα στείλετε μια επιστολή και στην περιφέρεια. Ναι, αυτό είναι το πρώτο που θα κάνουμε, λέει η Πρόεδρο. Θα διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά, θα στείλουμε μια επιστολή στην περιφέρεια και αν θέλετε μπορούμε να στείλουμε και μια επιστολή στην ΕΜΒΗ. Όχι αναγκαίο βέβαια αυτή τη στιγμή, ούτω ή άλλω θα κάνουμε ένα απολογισμό των όσων έχουμε, θα ξεκινήσουμε μια μελέτη και μετά βλέπουμε. Αλλά πρώτα απ' όλα να συζητηθεί μεταξύ συντονιστών. Ευχαριστώ. Ωραία, πολύ καλά. Καλή επιστροφή στην πανέμορφη περιοχή του Μιλάνου. Και συνεχίζουμε. Και περνάμε στο σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την αναφορά 0502, 0503 και 0506. Ο Κορνέλ Μπαλόγκε είναι ο αναφέρον για την 503. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πέντε λεπτά το πολύ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω βοήθεια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΜΣΜΑ. Είμαι ένα από τα θύματα τους Ούγκρους και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι η Iron FX αρνείται να αποσμιώσει τους πελάτες της. Εγώ είμαι ένας μικρός επενδυτής και δεν έχω ούτε τεράστια κέρδη, ούτε τεράστια απώλειες. Απλώς θέλω τα χρήματα τα οποία έχω βάλει στην πάντα για την οικογένειά μου να μπορέσω να το πάρω πίσω. Ποια είναι λοιπόν τώρα η κατάσταση. Θα συνοψίσω. Κάπου 1.700 μικροί επενδυτές ε, χρησιμοποίησαν ως ε, μεσαιτία συναλλάγματος την Iron FX. Είναι απίστευτο, αλλά η εταιρεία αυτή αρνείται να μας πληρώσει, να μας επιστρέψει τις καταθέσεις μας. Πάνω από 25.000 ευρώ έχω καταθέσει στην εταιρεία αυτή και ζήτησα να αποσύρω πριν από 20 μήνες και κάτι, δύο χρόνια δηλαδή περίπου τώρα, περιμένω για να πάρω πίσω τι, τα δικά μου τα χρήματα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αυτή η απάτη οφείλεται στην υπερβολική ελευθερία της αγοράς. Που σημαίνει ότι οι εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στην Κύπρο βρίσκονται υπό την εποπτεία μόνο των Κυπριακών αρχών. Έτσι όπως έχει σήμερα η κατάσταση, οι εποπτικές αρχές των ε, υπόλοιπων χωρών δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για τις επενδύσεις που βρίσκονται σε Κυπριακή έδρα. Δεν χρησιμοποίησε όμως ούτε η Επιτροπή Κεφαλαιογορών της Κύπρου τις εξουσίες της για να αλλάξει την κατάσταση. Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα και η εποπτεία, όπως είπαμε, είναι στην Επιτροπή αγορά Κύπρου. Δεν μπόρεσαν όμως να κάνουν την εποπτεία όπως πρέπει και έτσι η επενδυτική εταιρεία αυτή μπορεί ατιμωρητή να δράσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας την έδρα της στην Κύπρο. Αυτό έγινε με την Iron FX, η οποία αρνείται να πληρώνει πολλά εκατομμύρια στους πελάτες της και εξακολουθεί να έχει άδεια όμως και να μπορεί να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη. Αυτή η περίπτωση δείχνει πως οι εποπτικές κυπριακές αρχές παραβιάζουν τις αρχές της οδηγίας για τα μέσα των αγορών, τη MIFID δηλαδή, την οδηγία MIFID. Η Iron FX Global δεν συμμορφώνεται για μήνες τώρα με τις υποχρεώσεις της, έτσι όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 της οδηγίας MIFID. Με αποτέλεσμα να ζημιώνονται οι πελάτες. Δεν πρόκειται απλώς και μόνο για αμέλεια. Αυτά αναφέρονται και σε εκθέσεις της αρχής της Κύπρου. Η Iron FX λοιπόν Global φάνηκε ότι δεν έχει αρκετά χρήματα 176 εκατομμύρια λιγότερα δηλαδή που δεν μπορούσε να επιστρέψει στους πελάτες της και εξακολουθεί να μην μπορεί να τα επιστρέψει. Βάσει των στοιχείων αυτών, το άρθρο 8 της οδηγίας MIFID σύμφωνα με αυτήν θα έπρεπε οι αρχές της Κύπρου να αφαιρέσουν την άδεια από την επιχείρηση αυτή, γιατί η επιχείρηση δεν ανταπακρίνεται στις απαιτήσει οι οποίες είναι αναγκαίες για να μπορεί να έχει την άδεια. Επίσης υπάρχει και θέμα μη συμμόρφωσης των αρχών ασφάλειας αγορών της Ευρωπαϊκής Τέτοιας Αρχής. Στις 17 Μαρτίου Μαρτίου λοιπόν στείλαμε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Επιτροπή απάντησε ότι δεν μπορεί να ερευνήσει την υπόθεση αυτή της Iron FX. Όμως η αρχή κεφαλαίου μπορεί να κάνει τέτοια έρευνα και μάλιστα να απευθυνθεί και στις ίδιες τις ε, μεσαιτήσεις συναλλάγματος. Βάσει του άρθρου 17 τώρα της ΕΣΜΑ, έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει έρευνες. Οπότε αναρωτιέμαι γιατί δεν το κάνουν και γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει καμιά έρευνα που γίνεται. Είναι μεγάλος αριθμός των ε, πολιτών που απευθύνθηκαν στην ΕΣΜΑ, χωρίς όμως η ΕΣΜΑ να κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει διαφάνεια λοιπόν από τις ευρωπαϊκές αρχές. Και υπάρχει ατιμορρησία και γιατί υπάρχει ατιμορρησία, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια από τις κυπριακές και ευρωπαϊκές αρχές. Ο καταναλωτή δεν ξέρει κατά πόσον οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν προχωρήσει σε έρευνες κατά τέτοιων απατών. Οπότε είμαι και εγώ πελάτης, οι πελάτες διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει διαφάνεια γιατί κάθε φορά που διαμαρτύρονται στις ευρωπαϊκές αρχές αυτό διαπιστώνουν. Θέλω λοιπόν απλώς να ζητήσω τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας προς τους μικρούς επενδυτές οι οποίοι έδειξαν εμπιστοσύνη στους ρυθμιστές και πίστεψαν ότι και οι Iron FX θα συμμορφώνονταν. Δεν ξέρω πια τι να κάνω. Πολλοί κόσμος φοβάται για την κατάσταση αυτή. Είναι απελπισμένοι. Εσείς είσαστε η τελευταία ελπίδα που μπορούν να έχουν οι οικογένειες αυτών των μικρών επενδυτών. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι έχουμε και άλλους ε, αναφέροντες οι οποίοι παρακολουθούν στο διαδίκτυο την συνεδρίασή μας, οπότε παρακολούθησαν και την παρουσία σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα να απαντήσει. Παρακαλώ, ο κύριος Αντρίτσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά τις τρεις αυτές αναφορές που συζητάμε, 502, 503 και 506 του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει γνώση πολυάριθμων καταγγελιών που έχουν υποβληθεί σε σχέση με εικαζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και πιο συγκεκριμένα για την Iron FX εταιρεία επενδύσεων με έδρα την Κύπρο που από τους ρυθμιστές, του Κύπριους. Όπως είπε και ο με τους σημερινούς κανόνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εξουσίες για να παρέμβει σε ατομικές περιπτώσεις. Η επιβολή των ε, κανόνων είναι ευθύνη των εθνικών ρυθμιστών που έχουν βέβαια και το καθήκον να εποπτεύουν τις αγορές και να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες. Όσον αφορά λοιπόν τώρα τα παράπονα που έχουν υποβληθεί για την Iron FX, είναι ο Εθνικός Εθμιστής της Κύπρου και τα Κυπριακά Δικαστήρια, τα οποία θα ερευνήσουν αν υπήρξαν παραβιάσεις, όπως στην περίπτωση αυτή για την Iron FX, ή στην νομοθεσία, αν δεν μετέφερε καλά στην εθνική νομοθεσία τους ευρωπαϊκούς νόμους. Θα δώσω τώρα το λόγο και στον κύριο Ντέκερ από την ε, Τιτζιτζάς Just της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα σας πει περισσότερα. Ευχαριστώ και εγώ και σας ευχαριστώ όλους. Κύριε Πρόεδρε, παρεμβαίνω για να αναφέρω κάτι το οποίο δεν ακούστηκε από τον αναφέροντα, αλλά αναφέρεται στις τρεις αναφορές που εξετάζουμε σήμερα. Και αυτό έχει να κάνει με τις δικαστικές διαδικασίες οι οποίες έλαβαν ε, χώρα ε, με τον Ombudsman στην Κύπρο. Οι αναφορές λένε ότι δεν ικανοποιήθηκαν οι αναφέροντες κυρίως εξαιτίας της διάρκειας που κράτησαν οι δικαστικές διαδικασίες και για το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές. Και ότι πιθανότατα υπάρχει παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις εξώδικες ε, επιλύσεις διαφορών. Πρόκειται για την οδηγία 213 καθετός 11 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιπτώσεις αυτές εναλλακτική επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Η οδηγία 213-11 μιλάει για απαιτήσει ποιότητα όταν πρόκειται για τέτοιε διαδικασίε εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Και το πεδίο εφαρμογή τη περιορίζεται σε συγκεκριμένους οντότητες που έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει αυτής της οδηγίας. Το σύστημα δηλαδή που προβλέπεται από την οδηγία είναι ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν ε, πρόσβαση στις διαφορές που έχουν τις καταναλωτικές, να έχουν πρόσβαση λοιπόν στις, στους φορείς εναλλακτική επίλυσης, ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και ότι οι χώρες μέλη επιτρέπουν την πρόσβαση αυτή, ορίζοντας ποιοι είναι οι φορείς οι οποίοι μπορούν να δράσουν σε τέτοιες περιπτώσεις εναλλακτική επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Η Κύπρος έχει μια τέτοια, ένα τέτοιο φορέα που είναι η υπηρεσία προστασίας των καταναλωτών. Όπως είπα, οι απαιτήσει ποιότητας της οδηγίας περιλαμβάνουν και την απέτηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, δηλαδή την αναγκαιότητα μέσα σε 90 μέρες να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και αυτό έχει να κάνει μόνο με τις καταχωρημένες, τους καταχωρημένους φορείς. Η Κύπρος, όπως σας είπα, έχει καταχωρήσει ένα τέτοιο φορέα. Όχι όμως και στα πλαίσια του Ombudsman της Κύπρου. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε δυσαρέσκεια των αναφερόντων σχετικά με διαδικασίες ενώπιον του οικονομικού Ombudsman δεν μπορούν να προφασιστούν παραβίαση της οδηγίας 213 EU. Και θέλω να προσθέσω εδώ κυρία Πρόεδρε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην συνήθη άσκηση καθηκόντων της ελέγχων για την οδηγία αυτή εντοπίζει περιπτώσεις νομοθεσίας που εφαρμόζει η Κύπρος και έχουν υπάρξει διαδικασίες με πολύ καλή συνεργασία όμως ανάμεσα στην Επιτροπή και την Κύπρο επ' αυτών. Τώρα έχει εγκριθεί πολύ πρόσφατα νέα νομοθεσία, δημοσιοποιήθηκε την 7η Ιουλίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει για να δει κατά πόσο συμμορφώνεται όντως πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τόσα πολλά ζητήματα προκύπτουν. Ωραία. Οι συνάδελφοι θα πάρουν το λόγο σε λίγο. Πρώτα, η κυρία Βερλέο Ντανιάκ, που είναι η εκπρόσωπος της ΕΣΜΑ για την συμμόρφωση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για αυτή την πρόσκληση. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει σοβαρά την ΕΣΜΑ τα τελευταία δύο έτη. Έχουμε δηλαδή λάβει καταγγελίες από κατανοητές από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης έχουν αναφερθεί και ανησυχίες από τις εποπτικές αρχές διαφόρων χρόνων, Οπότε ε, είναι σημαντικό να διερευνηθεί αυτό το ζήτημα προκειμένου να κατανοήσουμε και ποιος ακριβώς δικαιούται να κάνει τι στο σημερινό νομικό πλαίσιο. Ε, καταρχήν ε, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ήταν οι θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε δηλαδή η ΕΣΜΑ είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχουν το δικαίωμα να ε, επεμβαίνουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Δηλαδή οι αρμόδιες θεσμικές εθνικές αρχές, οι Επιτροπές Κεφαλαγοράς είναι εκείνες οι οποίες είναι αρμόδιες για την εποπτεία ε, και την εφαρμογή τη νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις εν λόγω επιχειρήσεις όπως οι Άρων FX που εμπίπτουν δηλαδή στη δικαιοδοσία τους. Ε, και ε, τελικά ο διαμεσολαβητής της Κύπρου και τα κυπριακά δικαστήρια είναι εκείνα που είναι σε τελική ανάλυση αρμόδια για την επίλυση διαφορών ε, μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων εδώ ε, Iron FX. Τώρα, γιατί ενδιαφέρει την ΕΣΜΑ αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, αυτή η υπόθεση, γιατί ε, κατά τελευταία δύο έτη λάβαμε 500 καταγγελίες μεμονωμένες ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, παράβαση, την άποψή του από την πλευρά τη Iron FX των διατάξεων τη ε, οδηγία MIFID. Και βέβαια όχι μόνο από την πλευρά τη Iron FX και εν λόγω καταγγελίε τελικά μετατράπηκαν σε καταγγελίε κατά της Επιτροπής Κεφαλακοράς, τη δυσμηθική δηλαδή αρχή της Κύπρου, επειδή δεν ανέλαβε δράση εδώ. Και σα είπα ότι υπάρχουν και μία σειρά από περαιτέρω ε, ρυθμιστικές εποπτικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που στράφηκαν στην ε, ΕΣΜΑ ε, επειδή ανέφεραν ότι υπάρχει ακριβώς παράβαση από όχι μόνο την πλευρά της Iron FX αλλά και από άλλες επιχειρήσεις που εδράζουν στην Κύπρο και οι οποίες εφαρμόζουν επιθετικές πολιτικές σε ό,τι αφορά την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της. Άρα λοιπόν η ΕΣΜΑ είναι αρμόδια για την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και ε, οφείλει να συμβάλλει στην συνεκτική και αποτελεσματική εποπτεία που ασκείται από την πλευρά των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Τι έχουμε λοιπόν κάνει εμείς από την πλευρά τη ε, ΕΣΜΑ. Εξετάσαμε το εν λόγω ζήτημα από τρεις οπτικέ γωνίε. Ε, καταρχήν συστάθηκε μια κοινή ομάδα εποπτών τον Ιούλιο του 2015 όπου περιλαμβάνονται εκπρόσωποι από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς της Κύπρου και από και άλλοι host supervisors από κράτη-μέλη. Και ε, εδώ ε, επικεφαλής ήταν ο διευθυντής της ΕΣΜΑ ε, προκειμένου να ε, υπάρξει εποπτεία των συγκεκριμένων δράσεων. Και αυτό ακολούθησε μετά η επιτόπια ε, ε, επιθεώρηση επιχειρήσεων οι οποίες ασκούν τη δραστηριότητά τους στην Κύπρο το 2015 και κατέληξε σε 8 κυρώσεις, δηλαδή επιβολή 8 κυρώσεων και μία ανάκληση άδεια ε, ασκησή δραστηριότητα. Ε, και ε, μία από τι επιχειρήσει στι οποίε επιβλήθηκε πρόστιμο ήταν η Iron FX και 2 εκατομμύρια ευρώ ήταν συνολικά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν. Από εκεί και μετά προβήκαμε στον έλεγχο 11 περαιτέρω επιχειρήσεων για τις οποίες υπήρχε υπόνοια σε ό,τι αφορά την ε, υπονόμευση της προστασίας των επενδυτών. Άρα λοιπόν εμείς εξετάσαμε από την πλευρά του επόπτη ως επόπτης ε, αυτό το ζήτημα λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ε, έχοντας κατά νου τη μόνη αρμόδια για την εποπτεία σε αυτή την περίπτωση είναι η Επιτροπή Κεφαλαγοράς της Κύπρου. Ε, προσπαθήσαμε όμως να, να διασφαλίσουμε ότι ακριβώ προβαίνει στην κατάλληλη παρακολούθηση και υποπτία ε, των δράσεων της Aronefex. Τώρα, δεύτερη οπτική γωνία είναι η κανονιστικού χαρακτήρα. Εκεί δημιουργήθηκε λοιπόν μια task force από την πλευρά τη ΕΣΜΑ, η οποία περιλαμβάνει μέλη από όλε τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατομελών τη της Ευρωπαϊκής προκειμένου να εξεταστούν αυτά τα περίπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα, στα οποία ε, περιλαμβάνονται τα contract for differences, CFTs, αλλά και ε, ε, άλλα προθεσμιακά προϊόντα. Ε, υπήρξαν εκεί ε, δύο έγγραφα, ε, ένα έγγραφο Q&A και δύο περαιτέρω έγγραφα, το τελευταίο από αυτά τον Ιούλιο του 2016, στο οποίο αναφέρουμε ξεκάθαρα ότι τα λόγο προϊόντα είναι επικίνδυνα και δεν θα πρέπει να παρέχονται χωρίς να έχει υπάρξει κατάλληλη παροχή συμβουλών στους επενδυτές αφού μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες ζημίες. Επίσης, εκεί αναφέρουμε ότι η ΕΣΜΑ εξετάζει ε, τον τρόπο με τον οποίο ε, θα μπορεί να ασκεί ε, με τον καλύτερο τρόπο της αρμοδιότητας της από τον Ιανουάριο του 2018 στα πλαίσια δηλαδή της εφαρμογής της νέας οδηγίας MIFID 2. Από εκεί και μετά υπήρξε μια πολυμερής δράση από την ΕΣΜΑ και, της, και την και σε ό,τι αφορά αιτήματα για παροχή πληροφοριών τόσο από την πλευρά τη ε, Επιτροπή και τη Κύπρου, όσο και από την πλευρά τη ε, ΕΣΜΑ, προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω διευκρινήσει σε ό,τι αφορά ε, την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή τη Κύπρου. Η εν λόγω βέβαια αλληλογραφία ήταν και παραμένει εμπιστευτικού χαρακτήρα, οπότε θα περιοριστώ εδώ. Όμως, τα όσα κάναμε στο πλαίσιο αυτής της αλλαγογραφίας σε συνεργασία με τα όσα έκανε και η μικρή ομάδα εργασίας ε, μπορεί να επιτρέψει στην ΕΣΜΑ να αποφασίσει ε, το κατά πόσο μπορεί να ε, ξεκινήσει μια επίσημη διαδικασία και κατά πόσο θα είναι ε, επαρκή σε κατάλληλη αυτή η διαδικασία στο πλαίσιο δηλαδή της εφαρμογής του άρθρου 17 σε ό,τι αφορά παραβίαση ενωσιακής νομοθεσίας. Άρα λοιπόν, εδώ υπενθυμίζω ότι ε, σε ό,τι αφορά αυτήν την, ε, την εφαρμογή του άρθρου 17 έχουμε να κάνουμε με ζήτημα αρμοδιότητας της ΕΣΜΑ. Και για να ληφθεί η σχετική απόφαση η ΕΣΜΑ ελαμβάνει υπόψη της και το τι μπορεί να αναμένει ως αποτέλεσμα από μια επίσημη τέτοια έρευνα, ε, συμπληρωματικά δηλαδή στα όσα προέκυψαν ε, κατά τα τελευταία δύο έτη. Εάν συμφωνήσει τελικά το Διοικητικό Συμβούλιο και υπάρξει μια επίσημη διαρεύνηση, θα υπάρξει μια επίσημη ε, σύσταση από το τη ΕΣΜΑ. Τώρα, εάν η Επιτροπή υιοθετήσει αυτή την ε, γνωμοδότηση, τότε θα έχουμε να κάνουμε μια επίσημη γνωμοδότηση από πλευρά τη Επιτροπή πλέον και όχι τη ΕΣΜΑ. Αλλά αυτό που. Ε, ενδεχομένω να μην κατάλαβε καλά ο κύριο Βαλούν, είναι ότι ε, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπάρξει μια συγκεκριμένη γνωμοδότηση από πλευρά τη ΕΣΜΑ σε ό,τι αφορά την Iron FX. Γιατί όπω βλέπει στο άρθρο 17, ε, παράγραφο 6, μια τέτοια δυνατότητα υπάρχει μόνο όταν έχουμε ε, διατάξει οι οποίε ισχύουν άμεσα απευθεία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά αυτό δεν, δεν συντρέχει εδώ γιατί ακριβώ δεν έχουμε να κάνουμε με κανονισμό αλλά με οδηγία ένα ε, τέτοιο ε, πάντως αίτημα σε ό,τι αφορά την επίσημη διεξαγωγή, τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας από την ε, ΕΣΜΑ δεν έχει ληφθεί ακόμα. Εμείς θέλαμε καταρχήν να ε, δούμε τι ακριβώς έχει διερευνήσει η Επιτροπή Κεφαλαγόρας της Κύπρου και μια απόφαση για την έναρξη επίσημης έρευνας θα ληφθεί το φθινόπωρο. Τέλος να σας πω ότι ε, από την πλευρά της ΕΣΜΑ πάντοτε απαντήσαμε σε όλες τις καταγγελίες τις οποίες λάβαμε παρά τον τεράστιο αριθμό τους, όπως σας είπα 500 καταγγελίες που βέβαια οδήγησαν ε, σε περαιτέρω αλληλογραφία, εκτεταμένη αλληλογραφία με την ε, ΕΣΜΑ. Ε, και πάντοτε εμείς ε, βαίνουμε και σε περαιτέρω ε, ενημέρωση των καταγγελόντων, εντάξει όχι κάθε δύο εβδομάδες, αλλά εντός έξι μηνών πάντοτε σε ό,τι αφορά δηλαδή και την αξιολόγηση των περαιτέρω μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν. Περιορίζομαι σε αυτά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε. Ήταν πολύ σαφή. Ευχαριστούμε που προσπαθήσατε να μας εξηγήσετε την κατάσταση και την πολυπλοκότητά της δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πώς συνέβησαν όλα αυτά. Έχω πολλές ερωτήσεις και εγώ ίδια, αλλά θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Παπαδάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω λάβει σχετική πληροφόρηση μετά από τις ε, καταγγελίες των παραπονωμένων και αυτό το οποίο γνωρίζω αυτή τη στιγμή είναι ότι η υπόθεση βρίσκεται στο χρηματοοικονομικό νόμπουσμα όπου ε, θα πάρει την απόφαση, δεν έχει εξεταστεί μέχρι σήμερα η όλη υπόθεση και αν αποφασίσει ότι οι παραπονούμενοι έχουν δίκιο θα πρέπει η άμεσα η εταιρεία να τους αποζημιώσει. Αυτό, αυτά έχουν έρθει, περιέρθει στη δική μου αντίληψη μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Can also add some... Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ κάποια ερωτήματα. Εάν δεν υπάρχει προστασία, η πανευρωπαϊκή προστασία που όπως φαίνεται ισχύει τελικά για πολλές, για εκατοντάδες υποθέσεις και φαίνεται ότι η ΕΣΜΑ είναι τόσο δημοφιλής όσο και η Επιτροπή Αναφορών. Τόσες πολλές επιστολές λαμβάνει. Έχουμε πολλές ομοιότητες λοιπόν έτσι. Για ποιο το λόγο λοιπόν επιτρέπεται η συναλλαγή με τέτοιες ε, ύποπτες εταιρείε. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται εύλογα. Και δεύτερον, γιατί οι υποθέσεις αυτές ε, αντιμετωπίζονται ε, μία προς μία, ενώ είναι χιλιάδες. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια δυνατότητα συλλογικής αποκατάστασης. Αυτό θα ήταν το φυσιολογικό. Και τρίτον, έχετε ήδη επιβάλει κυρώσεις σε ορισμένες επιχειρήσεις, προειδοποιήσεις τι αναμένεται να γίνει, μπορεί να ανακληθούν τα δικαιώματά τους, οι αδειές τους τέτοιων εταιριών που λειτουργούν εντελώς αδιαφανώς, για να μην πω χειρότερα. Υπάρχει κάποιος από εσάς που θα ήθελε να απαντήσει, η Κομισιόν ενδεχομένω, η ΕΣΜΑ. Shall I start? Um, Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ε, χρειάζεται ομαδική προσπάθεια εδώ για να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις. Ε, να ξεκινήσω με τη δική σας ερώτηση. Ε, γιατί επιτρέπονται οι συναλλαγές Εκεί πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχική μου παρέμβαση ότι εξαρτάται από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή να παρέμβει, να επαληθεύσει εάν η επιχείρηση που παρέχει τέτοια προϊόντα είναι ε, λειτουργεί ορθά ε, και εντός των ορίων ε, της νομότητας. Τώρα, όσον αφορά την κατά περίπτωση αντιμετώπιση, ο ρόλος της Κομισιόν όσον αφορά τη μεταφορά μιας οδηγίας είναι να ο να ελέγχει ότι οι κανόνες έχουν μεταφερθεί σωστά, με ακρίβεια από τα κράτη-μέλη και σε αυτή την περίπτωση από την Κύπρο. Η Κομισιόν μπορεί να παρέμβει αν διαπιστώσει ότι η μεταφορά των κανόνων δεν έγινε σωστά. Ωστόσο, κοιτώντας ε, τις καταγγελίες εδώ, αφορούν μια επενδυτική εταιρεία χωρίς να αναφέρεται οποιαδήποτε, οποιοδήποτε οριζόντιο λάθος, συστημικό λάθος, ε, συστημική ανακριβής μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Γι' αυτό το λόγο οι καταγγελίες αυτές αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Όσον αφορά την ερώτηση για τον Σολαβήτη, ο συνάδελφός μου θα μπορούσε να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, θέλετε να μάθετε γιατί δεν αντιμετωπίζουμε συλλογικά όλες αυτές τις υποθέσεις. Ε, αν το δούμε από την πλευρά του πλαισίου εναλλακτική επίλυση διαφορών, τίποτα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν ε, εμποδίζει τα κράτη-μέλη να επιλέξουν το σύστημα που θέλουν να δημιουργήσουν. Μπορούν να έχουν λοιπόν και συστήματα εναλλακτική επίλυση διαφορών που θα επιτρέπουν συλλογικέ διαδικασίε, αλλά μπορούν να επιλέξουν, όπω είναι συμβαίνει, συγκεκριμένους ε, οργανισμούς που ασχολούνται με επιμέρους ε, ε, υποθέσεις διαφορών. Όσον αφορά τη δικαστική αποκατάσταση, τα... θα ξέρετε ότι υπάρχει μια σύσταση της Επιτροπής του 2013 για τα συλλογικά ένδικα μέσα που συνιστά στα κράτη-μέλη που δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να προσφέρουν ενδικά μέσα για διαφορές και τέτοιου είδους σαν αυτές που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Η σύσταση αυτή ε, προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά, συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες και η Κομισιόν αξιολογεί της συστάσεις του 2013 Εντό δύο ετών τα κράτη-μέλη πρέπει να εξετάζουν το ζήτημα και μετά από άλλα δύο χρόνια η Κομισιόν αξιολογεί το τι έχει γίνει οπότε η άσκηση αυτή ουσιαστικά θα γίνει φέτος από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Μία απάντηση φυσικά είναι ότι προφανώς έχουμε να κάνουμε με οδηγίες και όχι κανονισμούς και αν ε, δεν είσαι τυχερός επενδύεις στη λάθος χώρα. Έτσι έχουν τα πράγματα να ξαναδώσω το λόγο στον αναφέροντα για άλλα δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ε, πρέπει να πω πως απευθύνθηκα σε όλες τις αρχές, δηλαδή απευθύνθηκα και στο νομικό ομπουτσμαν και στην Επιτροπή Κεφαλαγοράς της Κύπρου και θα πρέπει να πω ότι η Επιτροπή Κεφαλαγοράς ούτε καν απάντησε στην καταγγελία μου, ενώ η υπόθεση ενώπιον του ομπουτσμαν ε, τρέχει εδώ και ε, 20 μήνες. Άρα λοιπόν ο χρηματοοικονομικό επίτροπο στην ε, διαμεσολαβητή συγγνώμη δεν έχει κάποια προθεσμία που να το δεσμεύει, οπότε η ολόκληρη διαδικασία ενώπιον του μπορεί να τρέξει ε, πάπυρον. οπότε και ακριβώ επειδή δεσμεύεται από κάποιο κανόνα δεν χρειάζεται να τηρήσει κάποιο όριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την, ε, την ΕΣΜΑ, στράφηκα στην ΕΣΜΑ, αλλά δεν ήταν σε θέση να κάνει κάτι για να με βοηθήσει. Οπότε το ερώτημα που θέτω είναι πού θα λάβουμε, από πού θα λάβουμε βοήθεια ως επενδυτές. Μπορώ προφανώς να ε, παράσχω τεκμήρια, να παράσχω δικαιολογητικά έγγραφα, έχω τα πάντα στη διάθεσή μου, αριθμούς αναφοράς και ούτω καθεξής. Αλλά ε, ε, πρέπει να πω ότι διαφωνώ με τη δήλωση της ΕΣΜΑ ως προς το ότι ε, δεν είναι αρμόδια ε, για την ε, επίλυση διαφορών σε ό,τι αφορά δηλαδή μονομένες υποθέσεις. Όμως στην περίπτωση της Κύπρου έχουμε ε, την Κύπρο ως μια χώρα στην οποία ε, έχουν την έδρα τους 228, 228 ε, επενδυτικές εταιρείες χωρίς όμως να, έχουν, να έχει δημιουργήσει τα κατάλληλα εργαλεία για την προστασία των επενδυτών. Δεν έχει για παράδειγμα ένα ταμείο αποθεματικό σε ό,τι αφορά την προστασία των επενδυτών, δεν έχει εφαρμόσει άλλες και θα πρέπει να πω ότι αυτές οι επιχειρήσεις επενδυτικές δηλαδή, οι 228 που έχουν την έδρα τους στην Κύπρο, έχουν τη δυνατότητα να ασκούν δραστηριότητα στην ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, παγόμενες όμως την εποπτεία ε, της Επιτροπής Κεφαλαγοράς της Κύπρου και χωρίς να ξέρουμε αν τελικά αυτή η έλλειψη εποπτείας είναι αποτέλεσμα αναποτελεσματικότητας ή διαφθοράς. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρο. Λαμβάνουμε υπόψη μα αυτά τα σχόλια που κάνατε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να συνοψίσουμε λέγοντα ότι θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά σα και θα ζητήσουμε μία ενημέρωση από την Επιτροπή, ειδικότερα σε ό,τι αφορά ε, το ζήτημα ε, της ε, ουσιαστικής προστασίας ε, και της έλλειψης διαφάνειας, αλλά και σε ό,τι αφορά το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαγορά της Κύπρου. Δηλαδή, αν έχει λίγο προσωπικό, λίγους υπαλλήλους και οι μισοί λείπουν σε άδεια και άλλοι μισοί έχουν ασθενήσει, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα εκεί ίσως θα μπορούσαμε να ε, ε, απευθύνουμε και μία επιστολή τόσο στην Επιτροπή Αγοράς όσο και στο χρηματοοικονομικό ομπουτσμαν της Κύπρου που αναφέρθηκε προκειμένου να εκφράσουμε την ανησυχία μας σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις, σε ό,τι αφορά την έλλειψη διαφάνειας και να ζητήσουμε την δική τους ε, συμβουλή ως προς τα επόμενα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Τέλος, πιστεύω ότι χωρί καμία καθυστέρηση θα πρέπει να στραφούμε στον Ευρωπαίο, στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και να τη ζητήσουν να μας πει γιατί δεν έχει γίνει ε, περαιτέρω διερεύνηση αυτής της υπόθεσης σε ό,τι αφορά ε, την ε, άσκηση, δηλαδή κατάλληλα υποπτήρια από την πλευρά της Επιτροπής Κεφαλαγοράς της Κύπρου απέναντι στην Ε, Δεν ξέρω αν συμφωνούν οι συνάδελφοι με τα όσα πρότεινα. Καλώς, έτσι θα προχωρήσουμε. Καλώς, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε κάποιον άλλον σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Οπότε πάμε στο επόμενο σημείο 1109 σε ό,τι αφορά τον ε, νέο ε, φόρο βιώσιμου τουρισμού στις Βαλεαρίδες νήσους. Ε, ο Μανουέλ Σαντίνο Λόπες, ο αναφέρον, είναι εδώ, βρίσκεται μαζί μας σήμερα, οπότε του δίνω το λόγο για 5 λεπτά. Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας που μας δίνετε την ευκαιρία να έρθουμε και να απευθυνθούμε στο σώμα. Θέλω να απαντήσω στα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπόθεση αυτή φαίνεται κατάσταση αλλιώ από την, γιατί η Επιτροπή δέχεται ότι η διάκριση μπορεί να υπάρχει. Εμείς λέμε ότι όντως υπάρχει. Επίσης η Επιτροπή μπερδεύει το ποια είναι η διάκριση. Γιατί η κυριαρχία της κυβέρνησης των Βαλαρίδων Ίσων περιορίζεται στις Βαλαρίδες Νήσους. Η διάκριση γίνεται ανάμεσα στους κατοίκους των Βαλαρίδων Νήσων και των υπολείπων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των Ισπανών που δεν κατοικούν όμως στις Βαλερίδες νήσους. Αυτοί που κατοικούν εκεί πληρώνουν 0,26% φόρο. Οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ισπανοί, που δεν ζουν όμως στις Βαλερίδες ε, νήσους, πληρώνουν το 93,5%. Οπότε, ναι, επίσημα όλοι πληρώνουμε τα ίδια. Κάτω από αυτή την κατάσταση, οι οικονομολόγοι τι λένε, λένε ότι πρόκειται για εξαγωγή φόρων. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι και καλυμμένη. Υπάρχουν και άρθρα στον τύπο που το αποδεικνύουν αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά κάτι παρόμοιο παρά μόνο στην Καταλωνία. Εμείς είμαστε μόνοι στην Ισπανία και στην Ευρώπη που έχουμε αυτή τη σύλληψη φόρου. Γιατί τελικά πληρώνει κανεί για την οικονομική ικανότητα που έχει να ταξιδέψει και να διαμείνει για κάποιο χρόνο στις Βαλερίδες νήσους. Και όσο πιο πολύ μένει, τόσο πιο φτηνό φόρο πληρώνει. Αυτό βέβαια είναι κάπως αντιφατικό. Επίσης, είναι περίεργα τα πράγματα γιατί πρόκειται και για κάτι περιφερειακό και όχι δημοτικό. Και είναι και μοναδική περίπτωση γιατί τελικά δεν πρόκειται για φόρους, αλλά μάλλον γιατί δεν πρόκειται για τέλη, αλλά πρόκειται για έναν φόρο. Καθαρά φόρο που δεν είναι όμως αντισταθμιστικός. Δεν ανταποκρίνεται σε κάποιες υπηρεσίες που δεχόμαστε. Για ποιο λόγο υπάρχει λοιπόν αυτή η διάκριση. Η Επιτροπή δίνει ε, παραδείγματα και λέει ότι να θα υπάρξουν υδροελεκτρικά έργα και ίσως γι' αυτό. Η ίδια όμως η κυβέρνηση που παίρνει τον τουριστικό αυτό φόρο συγχρόνως εφαρμόζει και ένα διάταγμα για την καθαρότητα των υδάτων και το πρώτο άρθρο λέει ότι χρησιμεύει για να πληρωθούν πολιτικές σχετικές με τα ύδατα στις βαλαρίδες νήσους. Δηλαδή εκεί τελικά πάει και ο φόρος από τους τουρίστες και προτιμά η κυβέρνηση των Βαλερίδων Ίσων να δημιουργήσει έναν άδικο φόρο για τους ξένους τουρίστες που έρχονται στις Βαλερίδες νήσους. Για μας ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι ξεκάθαρο. Όποιος πληρώνει το φόρο για το νερό είναι κάτοικος, μόνιμος. Ενώ ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν τελικά τον φόρο, τον τουριστικό, σχεδόν κανείς. ποιος ανακατεύεται σε όλα αυτά τα διάφορα τμήματα, περιβάλλον ε, κλπ. Δεν πρόκειται όμως καν για αντιστάθμιση από τη δραστηριότητα του τουρισμού. Και εδώ θα σας πω τι είπε ο ίδιος ο δικηγόρος της κυβέρνησης των Βαλαιορίδων για το φόρο αυτό. Λέει ότι πρόκειται για μία απόδοση καθαρά φορολογικού χαρακτήρα, δηλαδή αύξηση των εσόδων από μία πηγή πλούτου. Ο φόρος δεν μπορεί να θεωρηθεί νομικά σαν μία περιβαλλοντική απόδοση βάσει της αρχής οριπένων πληρώνει. Όλα αυτά τα είπε ο ίδιος ο δικηγόρος της κυβέρνησης των Βαλαριδονίστων. Δεν είναι λοιπόν φυσιολογικό. Πριν από μία εβδομάδα στη συνεδρίαση προέβλεψαν ένα διαγωνισμό ιδεών για να δουν πού τελικά θα πάνε τα χρήματα αυτά. Αν υπήρχαν ε, λόγια ανώτερη βία, δεν θα είχε νόημα να ψάχνουν πού θα ξοδέψουν τα χρήματα και όμως η κυβέρνηση ψάχνει να βρει τι θα τα κάνει αυτά τα χρήματα. Έπειτα πρόκειται για έναν φόρο που επιβάλλεται επιπλέον του ΦΠΑ. Δεν έχω χρόνο τώρα για να σας δώσω τις λεπτομέρειες. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ μένει στην επιφάνεια διότι πρόκειται για ένα φόρο ο έχει σχεδιαστεί για να δείχνει ότι δεν είναι όπως ο ΦΠΑ. Όμως δεν βρήκα κανέναν που να μπορεί να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην ε, παραμονή σε ξενοδοχείο που να τις επιβάλλει το ένας ή ο άλλος φόρος. Κανείς δεν μπορεί να κοιμηθεί σε ένα ξενοδοχείο χωρίς να πληρώσει και τους δύο φόρους. Άρα δεν πρόκειται για συσσόρευση φόρων, διπλή φορολόγηση. Η Ισπανία εφαρμόζει το άρθρο 78 της ε, οδηγίας για τον ΦΠΑ. Και τελειώνω ζητώντα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσει αυτή την υπόθεση με τους φόρους και να ζητήσει από το Βασίλειο της Ισπανίας να διορθώσει αυτή την κατάσταση που είναι άδικη για τους Ευρωπαίους τουρίστες. Αντίθετα με αυτά που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο έχουμε τεκμηρίωση στη διάθεσή μας και είμαστε και στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο θελήσετε να μας ρωτήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ο εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο κ. Μόλις Παλέχα, βρίσκεται εδώ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο φόρος αυτός τουριστικής ε, διαμονής επιβάλλεται στα ξενοδοχεία και άλλα καταλήματα τουριστικά σε κρουαζιερόπλια που σταματούν στις βαλερίδες νήσους και πρόκειται για έναν φόρο που δεν ε, κάνει διάκριση απευθείας στους ε, πολίτες που δεν είναι από την Ισπανία, γιατί πρόκειται και για κατοίκους και μη κατοίκου, για Ισπανούς, για μη Ισπανούς, άπαξ και αυτοί κατοικούν σε κάποιο ε, τουριστικό κατάλημα στις Βαλερίδες νήσους. Εκεί που υπάρχει διάκριση είναι έμεση. Όμως η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η έμεση διάκριση παρόλα αυτά δεν αποδεικνύεται. Για να υπάρχει έμεση διάκριση ένας φόρος πρέπει να έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που ακόμα και αν θεωρητικά επιβάλλεται εξάλλου στους ντόπιου και στους ξένους, στην πράξη επιβάλλεται μόνο στους ξένους. Και γι' αυτό ζητήσαμε στοιχεία στατιστικά για να δούμε ποιος φόρος επιβάλλεται παραπάνω στους μη κατοίκους. Ο φόρος αυτός όμως επιβάλλεται και σε Ισπανούς που κατοικούν εκτός Βαλερίδων ίσων. Στην πράξη λοιπόν, όπως είπε και ο αναφέρον, υπάρχουν στις χώρες μέλη και άλλοι τοπικοί περιφερειακοί φόροι που επιβάλλονται σε τουριστικά καταλήματα. Στην πράξη, πολλοί από αυτούς τους φόρους επιβάλλονται πιο συχνά στους μη κατοίκους τη συγκεκριμένη περιοχή Δήμου κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση των Βαλερίδων Ίσων, δεν αποτελούν εξαίρεση. Τώρα το γεγονός ότι επιβάλλεται πιο συχνά σε ξένους και όχι σε Ισπανούς, αυτό είναι συνέπεια του γεγονότος ότι οι Βαλερίδες νήσοι αποτελούν τουριστικό προορισμό, ιδιαίτερα δημοφιλή. Με αποτέλεσμα, πολλοί πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνουν, διαλέγουν για τις διακοπές τους τις βαλερίδες νήσους. Οπότε, μια απλή ποσοτική μελέτη πόσοι τουρίστες είναι ξένοι και πόσοι τουρίστες δεν κατοικούν στις βαλερίδες δεν φτάνει για να αποδειχτεί η έμεση αυτή διάκριση. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που θα μπορούσαμε να το αποδείξουμε κάτι τέτοιο. Εμεί πιστεύουμε ότι δεν αποδεικνύεται. Αλλά ακόμα και αν μπορούσε να αποδειχτεί ότι υπάρχει μια τέτοια διάκριση, μια που πρόκειται για ένα τέλος, σκοπός του οποίου είναι να δημιουργηθεί ένα ταμείο υπέρ προγραμμάτων για τον ε, βιώσιμο τουρισμό, θα έπρεπε κανείς να μελετήσει και να αναλύσει σε τι βαθμό η χρήση των κονδυλίων αυτών είναι κοινωνικού συμφέροντος ή οδηγεί σε μία διάκριση. Μέχρι τώρα η Επιτροπή εκτιμάει ότι δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Λέει η αναφορά ότι ο φόρος αυτός, το τέλος αυτό, αντιτίθεται, παραβιάζει την οδηγία για το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ όμως είναι συμβατός με άλλα τέλη, με άλλους ειδικούς φόρους. Όπως για τα καπνά, για τα νοπνευματόδη, για τις πινακίδες αυτοκινήτων. Οπότε θεωρούμε ότι το τέλος αυτό είναι συμβατό με τον ΦΠΑ. Τώρα αυτό είναι βέβαιο. Η οδηγία για το ΦΠΑ απαγορεύει στις χώρες μέλη το εξή. Να μην μπορεί μια χώρα να επιβάλλει ίδιο φόρο όπως είναι ο ΦΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η απέτηση. Το ΦΠΑ είναι ένας φόρος που επιβάλλεται σε όλα τα προϊόντα, είναι γενικός στην εκπαίδευση, στα τρόφιμα, σε όλες τις πτυχές των αγαθών και των υπηρεσιών. Είναι ένας φόρος, όμως αυτός τώρα για τον οποίο μιλάμε, που επιβάλλεται μόνο στις βαλερίδες νήσους και μόνο στα τουριστικά καταλήματα. Οπότε με τίποτα δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον ΦΠΑ. Ευχαριστούμε. Δίνουμε το λόγο σε συναδέλφους. Η πρώτα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον αναφέροντα που ήρθε εκ μέρους της οργάνωσης ξενοδοχών των Βαλερίδων Νήσων. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποστηρίξουμε, να μην υποστηρίξουμε το τέλος αυτό που επιβάλλεται. Γιατί είναι κάτι καθαρά περιφαριακό και το ίδιο το Κοινοβούλιο των Βαλαιορίδων απεφάνθη και το 2016 ενέκρινε το σχετικό κανονισμό κυβέρνηση των Βαλαιορίδων Ίσων. Το θέμα είναι τώρα να δούμε κατά πόσο φόρος αυτός που ισχύει είναι συμβατός με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Με πρώτη ματιά, από αυτά που είπε η Επιτροπή, εγώ θα έλεγα πως όχι. Από την ανταλλαγή. Οι ξενοδόχοι της Συμπίθα ζήτησαν από την Κομισιόν μία διευκρίνηση για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και η απάντηση που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι χωρίς να είναι βέβαιο 100% φαίνεται ότι δεν υπάρχει το σύμβατο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εγώ όταν πήγα στην Βήθα ζήτησα περισσότερα στοιχεία ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε μια απάντηση. Υπάρχει ή δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους ε, κατοίκους και τους μη κατοίκους. Πέρυσι το 2016. 26 Αυγούστου η ξενοδόχη της Βήθα ε, ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή απάντησε. Όμω η ξενοδόχοι τη Μαγιόρκα που έχουν τα ίδια συμφέροντα έκανε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα πήγε το τέλος αυτό στο δικαστήριο στις Βαλερίδες ε, νήσους, στο νότο δικαστήριο. Η διαδικασία άρχισε το 2016 και τώρα περιμένουμε την απάντηση του δικαστηρίου, του τοπικού. Έκανε όμω και κάτι άλλο η Μαγιόρκα. Στι 31 Μαρτίου φέτος έστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή Juncker, προκειμένου η Επιτροπή Juncker, έχοντας όλα τα στοιχεία που ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πει κατά πόσο παραβιάζεται ή όχι η ευρωπαϊκή νομοθεσία επειδή διαπιστώνεται διάκριση ανάμεσα στους κατοίκους και μη κατοίκους. Πέρα από όλα τα επιχειρήματα που δώσατε, διάβασα και τα κείμενα των ε, ξενοδόχων ε, της Μαγιόρκας. Όντως είναι όλα τα καταλήμματα τα τουριστικά ε, στα λιμάνια και αλλού, αλλά υπάρχουν όμως τα καταλήματα αυτά που επιβάλλουν το τέλος σε αυτούς που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά έρχονται από αλλού. Οπότε θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στους ξενοδόχους της Μαγιόρκας και να δώσει την ίδια απάντηση όπως και στην Ιμπίθα. Δηλαδή μετά όταν θα έχουμε την απάντησή σας γραπτά στην ε, Ομοσπονδία της Μαγιόρκα που συνοδεύεται από όλη την τεκμηρίωση που ζητήσατε τότε αφού έχουμε την απάντησή σας αυτή, τότε θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με την ε, αναφορά. Δηλαδή μέχρι να έχουμε την απάντησή σας, ζητάω να κρατηθεί ανοιχτή η αναφορά αυτή. Ο κύριος Τερικάβρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Με κάθε συμπάθεια. Με ξέπληξε. Είναι πρώτη φορά που κάποιος από ένα συγκεκριμένο μέρος από όπου έρχεται η αναφορά, κάνει αναφορά για να υποστηρίξει όχι τους δικούς του, αλλά τους ξένους. Όντω είναι η πρώτη φορά. Αυτό εντυπωσιάζει. Τώρα εγώ δεν καταλαβαίνω καθόλου την αναφορά πρέπει να σας πω. Δεν την καταλαβαίνω. Και γιατί. Γιατί το πρόβλημα για μένα είναι ο όρος διάκριση. Χρησιμοποιούμε τη λέξη διάκριση λες και οποιαδήποτε διαφορά είναι και διάκριση. Εντάξει, ξένοι που πάνε στην πάλμα της Μαγιόρκα μπορεί να έχουν άλλη διαφορά. Αυτοί που πάνε στην Καταλωνία, γιατί πάνε στην Καταλωνία κάποιοι, πάνε ή αυτοί που ζουν στη Μαδρίτη δεν πληρώνουν στους αυτοκινητοδρόμους διόδια. Στην Καταλωνία πληρώνουν. Είναι διάκριση αυτή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν ένα σωρό διαφορέ που δεν είναι απαραίτητα διάκριση. Ο όρος διάκριση είναι τόσο πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί που δεν μας βοηθάει στη συζήτηση. Βέβαια αυτά τα τέλη υπάρχουν κι αλλού. Στον Μπιλμπάο ήμουνα και πλήρωσα κι εγώ και δεν είναι στην Καταλωνία, πόσο ξέρω τουλάχιστον. Κι όμως πλήρωσα κι εγώ εκεί τέτοιο φόρο. Κι αλλού υπάρχει. Επίσης, εσείς λέτε ότι ο στόχος συλλογή του φόρου αυτού είναι για κάτι συγκεκριμένο, αλλά διαπιστώσατε ότι υπάρχει και άλλος φόρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό. Με αυτό για μένα δεν είναι επιχείρημα. Μια κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλούς και διαφορετικούς φόρους για να πετύχει ένα συγκεκριμένο σκοπό δεν απαγορεύεται. Οπότε ειλικρινά δεν βλέπω καθόλου να έχει έτσι δύναμη αυτή η αναφορά και η επιχειρηματολογία είναι τόσο μπερδεμένη που εγώ θα έλεγα να την κλείσουμε. Και οι ξένοι ή οι Καταλανοί, τέλος πάντων, πάμε στη μαγέρκα, ε, να κάνουμε, θα πληρώνουμε 2 ευρώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ειλικρινά πολύ. Τώρα, Πήρατε το λόγο πάνω από πέντε λεφτά, οπότε διστάζω να σας ξαναδώσω το λόγο. Θα το κάνω αν μου υποσχεθείτε ότι θα μιλήσετε λιγότερο από ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα επιμείνω στην έννοια της διάκρισης. Για μας είναι προφανής. Η διάκριση έχει να κάνει με την ίδια την έννοια. Δηλαδή βρίσκουμε έναν ένα τέλος το οποίο επιβάλλεται στους ξένους μόνο. Οπότε τελικά χρησιμοποιούνται χρήματα κάποιου που δεν ζει στις Βαλερίδες νήσους για τις Βαλερίδες νήσους. Και όταν ε, το 90% που σας είπα το πληρώνουν ε, οι ξένοι, για μας πρόκειται για διάκριση. Γιατί τελικά ο Ευρωπαίος τουρίστας πληρώνει το κόστος που αντιστοιχεί και στους ίδιους τους κατοίκους των Βαλερίδων Ιστών. Σίγουρα πρέπει να πληρώνουν φόρους οι τουρίστες και τους πληρώνουν, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να συνοψίσουμε τώρα και όπως σαφώς εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχει λόγος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει σε επαφή με την Ισπανία για το τέλος αυτό, δεδομένου ότι το σημερινό τέλος λέτε ότι εφαρμόζεται και στους ντόπιου και στους ξένους. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να την κλείσουμε. Δεν είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ξέρω ότι είσαι από τις ε, βαλερίδες νήσους Ρώσα, αλλά προσπάθησε να είσαι λίγο αμερόληπτη. Εντάξει, πολύ σύντομο παρακαλώ. Δεν είναι ότι παίρνω θέση για το κατά πόσο υπάρχει διάκριση δεν υπάρχει. Αυτό που λέω είναι ότι υπάρχει κάτι γραπτό από την Ομοσπονδία της Μαγιόρκα της 31ης Μαρτίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έπρεπε να απαντήσει η Επιτροπή θα έλεγα να μην είναι ανοιχτή η αναφορά μέχρι να μας απαντήσει γραπτά η Επιτροπή σε αυτή την επιστολή και τότε να την κλείσουμε. Αλλά αν δεν ξέρουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μην την κλείσουμε. Σήμερα το πρωί μίλησα με την Κομισιόν και είπε ότι σε ένα-δύο μήνες θα έχουν απαντήσει. Ας περιμένουμε λοιπόν την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ξέρουμε τι έχουν απαντήσουν στις ε, καταγγελίες της Μαγιόρκα που είναι ακριβώς ίδιες με εκείνες της Ιμπίσα. Έχουν στείλει όλη την τεκμηρίωση που τους έχετε ζητήσει από τη Μαγιόρκα. Δεν μπορεί να είναι κανείς πιο αντικειμενικός. Εγώ δεν λέω εδώ πέρα ποιος έχει δίκιο. Λέω να περιμένουμε την επίσημη απάντηση, τίποτα άλλο. Πρόεδρος, τέλεια. Θα ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει για την επιστολή αυτή και μετά θα χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία Β και θα την κλείσουμε τότε την αναφορά. Οπότε περιμένουμε να μας απαντήσετε γρήγορα, έτσι, να αντιδράσετε γρήγορα. Καλώς, ευχαριστούμε. Και τώρα το 22 έχει αναβληθεί. Οπότε είμαστε τώρα στην 1088 σχετικά με καζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων από τον νόμο των ΗΠΑ, Foreign Account Tax Compliance και τις εξοδαφικές επιπτώσεις της νομοθεσίας των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αναφέρον είναι κάποιος, το οποίο αρχικά είναι JR. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω σοφά το πεντάλεπτο που μου δίνετε ε, στην αναφορά περιγράφεται αναλυτικά η νομιμότητα της ΦΑΤΚΑ ε, ως πράξη συμμόρφωσης φορολογικής και παραβιάζει μάλιστα αυτή η πράξη τα άρθρα 8, 13 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύνδεξης ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πολλές άλλες νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία λογαριασμών πληρωμών και το άρθρο 55 του Γαλλικού Συντάγματος επίσης παραβιάζεται και άλλα. Δεν θα σας περιγράψω άλλο την αναφορά γιατί εξηγεί αυτά τα ζητήματα λεπτομερώς. Σας εξηγήσω πώς λειτουργεί η ΦΑΤΚΑ και τι επιπτώσει έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί κομμάτι διαφόρων εξοδαφικών νομοθεσιών των ΗΠΑ και επηρεάζει ε, άτομα, εταιρείε, ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τι οικονομίε μα. Ε, τέθηκε σε ισχύ το 2010 για να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή Αμερικανών πολιτών σε λογαριασμού offshore. Ε, αναφερόταν σε κατοίκους των ΗΠΑ που έκρυβαν χρήματα από την εφορία των ΗΠΑ στην Ελβετία. Σίγουρα αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Ωστόσο τελικά καταλήγει, είναι να αναγκάζει ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μη αμερικανικά να κάνουν αναφορά, να, να στέλνουν στοιχεία Αμερικανών πολιτών, ε, πελατών τους στην Αμερική. Είναι όμως πολύ ευρία και ανακριβής ε, ο, ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται ποιος είναι πολίτης των ΗΠΑ. Όλοι είδαμε το λύκο της Wall Street και τελικά την πληρώνουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι παρα πολίτε με διπλή υπηκότητα. Είμαι και εγώ ένα από του κατατύχει Αμερικάνου. Ε, ε, κατατύχει Αμερικανό, είναι ουσιαστικά ένα ξένο πολίτη ο οποίο ε, από λόγω των γονιών του ή για κάποιο άλλο κατατύχει έχει πάρει την υπηκότητα την Αμερικανική. Ακούτε και την προφορά μου. Δεν είμαι Αμερικανός, δεν έχω ζήσει ποτέ στη ΣΥΠΑ, δεν έχω σπουδάσει ποτέ εκεί, δεν έχω συγγενείς εκεί. Δεν έχω αριθμό κοινωνική ασφάλιση εκεί, δεν έχω ψηφίσει ποτέ σε εκλογέ. Η ιστορία μου είναι πολύ απλή. Ο πατέρα μου είναι Ιρλανδό, η μητέρα μου είναι Γαλλίδα. Ο πατέρα μου σπούδαζε στο Χάρβαρτ και εγώ γεννήθηκα σε αμερικανικό έδαφο. Μεταχώρησαν οι γονεί μου, ο πατέρα μου επέστρεψε στο Κέμπριτζ, η μητέρα μου προσπάθησε να μείνει στην Αμερική και απελάστηκε όταν ήμουν πέντε. Και πώ έγινε εγώ, απελάθηκα ουσιαστικά από την Αμερική. Αλλά Είχα γεννηθεί όμω σε αμερικανικό έδαφο το οποίο σημαίνει, χωρί να μπω σε πολλές λεπτομέρειες ε, για τα νομικά θέματα, υπάρχουν δύο μοναδικά χαρακτηριστικά στην αμερικανική νομοθεσία. Ε, αυστηρό δικαίωμα υπηκότητα λόγω γέννηση. Μόλι γεννηθεί κάποιος στην Αμερική, ε, παίρνει αυτόματα την αμερικανική ηθαγένεια. Για μένα είναι σαν, μια, σαν ένα μικρόβιο που έχω κολλήσει, μια κάποια ασθένεια από την κόλλησα. Ακούγεται αστείο, αλλά δεν είναι τόσο αστείο αν δείτε τι μα συμβαίνει. Το δεύτερο που συμβαίνει είναι ότι η Αμερική ε, έχει τη φορολόγηση ε, βάσει ηθαγένειας. Σε κάθε άλλη χώρα που σκέφτεται τον εαυτό της ε, η φορολογία βασίζεται στην κατοικία. Εάν δηλαδή λαμβάνει κάποιες υπηρεσίες από το κράτος τότε πληρώνει για αυτές τις υπηρεσίες. Αλλά στην Αμερική αυτό δεν συμβαίνει. Τι κάνουν οι Αμερικανοί λοιπόν όπως και η Ερυθρέα που είναι η μόνη άλλη χώρα στον κόσμο που κάνει αυτό ε, φορολογούν τους ανθρώπους βάσει υπηκότητας. Εφόσον γεννηθεί κανείς Αμερικάνος υπήκος, φορολογείται για την ηθαγένειά του ε, φόρου ζωή. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η ΙΠΑ και η Ερυθρέα είναι οι μόνες δύο χώρες στον κόσμο που εφαρμόζουν τέτοια πρακτική και έχουν επικριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ε, στο ψήφισμα 2023. Μάλλον έχουν επικρίνει τα Ηνωμένα Έθνη την Ερυθρέα, αλλά όχι τη ΣΥΠΑ. Καλό θα ήταν να επέκριναν και τη ΣΥΠΑ με τον ίδιο τρόπο. Και τι κάνει ο ΦΑΤΚΑ. Μέχρι τον ΦΑΤΚΑ οι ΙΠΑ δεν είχαν τρόπο να αστυνομεύσουν ε, τη φορολόγηση βάση ηθαγένειας. Δεν μπορούσαν. Το IRS τη ΣΥΠΑ, δεν μπορεί να απλώσει το χέρι του σε ξένες χώρες χωρίς ε, εντολή. Τι έκαναν λοιπόν οι Αμερικάνοι. Βρήκαν το ΦΑΤΚΑ. Και τι κάνει ο ΦΑΤΚΑ, δίνει τη δυνατότητα στην εφορία των ΗΠΑ να εφαρμόσει τη φορολόγησή της εκτός ε, συνόρων. Αναγκάζει λοιπόν ε, ε, υπηκόους των ΗΠΑ να δίνουν φορολογικά στοιχεία στην Αμερική ενώ εκεί. Βρήκαν ένα πολύ έξυπνο τρόπο. Ουσιαστικά ανάγκασαν ευρωπαϊκές διεθνείς τράπεζες να τους στέλνουν τα στοιχεία. Είπαν δηλαδή στα ευρωπαϊκά ιδρύματα θα βρείτε όποιον Αμερικανό έχετε, θα, οποιονδήποτε έχει γεννηθεί στη ΣΥΠΑ και θα μας στέλνετε τα στοιχεία. Όπως είπαμε λοιπόν, κατά τύχη υπήκοοι δεν έχουμε καμία σχέση με τη ΣΥΠΑ αλλά μας φορολογούν. Πολλοί μας λένε δεν πρέπει να φοβάστε, δεν υπάρχει διπλή φορολόγηση. Πράγματι εγώ είμαι ε, ξένος, έχω διπλή υπηκότητα, αλλά ε, κάποια πράγματα που κερδίζω στη Γαλλία μπορώ να τα πληρώσω να φορολογηθούν στην Αμερική. Υπάρχουν πολλές συνέπειες. Ε, ε, υπάρχουν ε, ποινές για διάφορα πράγματα, τρομακτικά πράγματα που εγώ γνωρίζω ως κατά τύχη Αμερικανός. Εν μεταξύ τα τέλη των Αμερικανών δικαιών είναι τεράστια και τελικά έτσι απορροφούν τεράστια ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ΕΠΑ και βγάζουν χρήματα από εμά. Αυτό συμβαίνει. Ουσιαστικά εμείς είμαστε οι ε, παρείες ε, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής ε, Μηχανίας, μας αρνούνται στεγαστικά δάνεια, μπλοκάρονται συντάξεις, ή συγγνώμη, αναλήψεις. Είναι τρομακτικά αυτά που συμβαίνουν. Πολλοί κόσμοι μας λέει, μα αφήστε, εγκαταλείψτε την ε, αμερικανική σας υπηκότητα, αλλά αυτό είναι αδύνατο για όλους τους λόγους που βλέπετε εδώ σε αυτήν την ε, διαφάνεια. Ε, κοστίζει ε, για να απαλλαχθεί κάποιος από την αμερικανική υπηκότητα 20 με 25 δολάρια. Ε, γνωρίζουν οι την ύπαρξή μας. Τα πράσινα βιβλία του Ομπάμα 2016-2017 προτείνουν αμνηστία για μας. Υπάρχει και μια ετήσια έκθεση στο Κογκρέσο του 2015, 16, 17 που αναγνωρίζει την τεράστια αδικία που επιβάλλεται σε εμά. Έχουμε και τους Democrats Abroad που θέλουν να συμπεριλάβουν την αμνηστία για μας στι τελευταίες ε, προεδρικές εκλογές ε, οι δημοκράτε κατα... μάχονται κατά τη ΦΑΤΚΑ. Το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε, εγώ μίλησα με έναν σημαντικό δικηγόρο του IRS, μα είπε ότι οι γνωρίζουν του κατατύχει Αμερικανού, αλλά καλούν δεν σα βλέπουν, διότι κερδίζουν ένα σωρό χρήματα από εσά και κανεί δεν πρέπει να σα υπερασπιστεί. Ακόμα και δηλαδή μεγάλοι δικηγόροι στην Αμερική μα λένε το ίδιο. Η Επιτροπή ε, η Κομισιόν ε, ζητά εντολή για να διαπραγματευτεί το ΦΑΤΚΑ και απορρίφθηκε. Ε, γιατί λένε ότι το ΦΑΤΚΑ είναι θέμα διμερές μεταξύ χωρών. Οπότε λένε εμείς νύπτουμε τα σχήρα μας. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Η Γαλλία ηγείται τώρα τη ε, μάχη και εγώ είμαι πολύ περήφανο. Υπάρχει μια έκθεση 150 σελίδων για του ε, νόμου αυτού τη Αμερική και πώ επηρεάζουν τη Γαλλία. Εδώ βλέπετε την αμνηστία των Democrats Abroad και αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Ουσιαστικά ξέρουμε ότι οι ΙΠΑ αρνούνται να συνυπογράψουν την CRS, ε, την φάτκα του ΟΣΑ. Ε, ουσιαστικά μετατρέπονται στις νες, ε, στην Ελβετία. Δισεκατομμύρια δολάρια εξάγονται ουσιαστικά από ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Αμερική. Πολύθηκε με την αμοιβαιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ σας είχαν υποσχεθεί ε, αμοιβαιότητα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν ε, αμοιβαιότητα η οποία έπρεπε να έχει ε, εφαρμοστεί μέχρι τα τέλη του περασμένου έτους. Αλλά ξέρουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να περάσει την Αμερική αμοιβαιότητα, θα την μπλοκάρει το Κογκρέσο. Οπότε υπήρχε μια υπόσχεση αμοιβαιότητα που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπογράψει τη ΦΑΤΚΑ, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να τηρηθεί. Έχουν ήδη καθυστερήσει στην εφαρμογή. Οπότε αυτό που ζητάω εγώ σήμερα εδώ είναι θέλουμε οι Κομισιόν, όπω έχουν παλιότερα ε, για χώρε όπω η Ελβετία και το Μονακό, να ζητήσουν από τα κράτη-μέλη να του δώσουν εντολή ώστε συλλογικά να επανεδιαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τη ΦΑΚΑ με την Αμερική ε, ισχυριζόμενοι ότι δεν τηρούν την υπόσχεση αμοιβαιότητα και ε, για να βρεθεί μια δίκαιη λύση και να εφαρμοστεί η αμνηστία των κατατέχει Αμερικανών που αναγνωρίζουν όλοι στην Αμερική ότι έχει ήδη καθυστερήσει. Συγγνώμη που ξεπέρασα το χρόνο μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Νίκολο Μπριλιώνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και καλησπέρα. Όσον αφορά την αναφορά αυτή, είναι ένα περίπλοκο θέμα, το ξέρουμε. Και εδώ είμαστε διάφορες γενικές διευθύνσεις που έχουμε έρθει για την αναφορά έχει να κάνει με πολλά ζητήματα. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην παραβίαση της ε, οδηγίας για την πληρωμή λογαριασμών. Στην αναφορά ο ισχυρισμός είναι ότι αυτοί οι Αμερικανοί που έχουν ε, αποτύχημα ε, γεννηθεί στην Αμερική φοβούνται ότι βάσει των συμφωνίων ΦΑΤΚΑ που έχουν υπογράψει οι χώρες μέλη ε, κινδυνεύουν από κυρώσεις. Εδώ πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με την οδηγία αυτή, Payment Accounts Directive, όταν πρόκειται για Ευρωπαίους καταναλωτές και έχουν πρόσβαση σε ένα ειδικό προϊόν το οποίο αναφέρεται στην οδηγία, δεν υπάρχει δυνατότητα διάκρισης εξαιτίας του τόπου κατοικίας ή της υπηκότητας. Παρά δηλαδή την απέτηση να συμμορφώνονται με την ΦΑΤΚΑ οι τράπεζες βάσει των διεθνών συμφωνιών, πιστεύουμε ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να αρνηθούν πρόσβαση στους καταναλωτές που μόνιμα κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε θα ερευνούσαμε τους λόγους και θέλουμε πληροφορίε αν υπάρχει κάποια παραβίαση για την οδηγία αυτή, την PAD, Payment Accounts Directive. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Η οδηγία άρχισε να ισχύει επίσημα 18 Σεπτεμβρίου του 2016. Και τώρα ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο τίθεται και σε εφαρμογή. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου πάλι. Αν έχετε πληροφορίες, τότε να μας τις στείλετε, γιατί εμείς δεν τις έχουμε. Πρόεδρος, μην μπούμε σε διάλογο, αλλά όντως ό,τι πληροφορίες έχετε να τις δώσετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ωραία, περνάμε στον επόμενο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Σιλ Μίλλερ. Ευχαριστώ. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη. Και έχω να κάνω με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία τους, κάτι το οποίο αναφέρει στην αναφορά του αναφέρον. Πράγματι, χώρες μέλη όταν δίνουν ε, στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει του ΦΑΤΚΑ πρέπει να τηρούν το κεκτημένο, το άρθρο 8 δηλαδή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και η μεταφορά αυτή προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται πληροφοριακά βάσει των, της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομενων 5946 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την οδηγια 9546. Κάτι το οποίο τόνισε ο αναφέρον είναι το εύρος των δεδομένων που ζητούν οι Ηνωμένε Πολιτείες βάσει του ΦΑΤΚΑ. Οι αρχές που εφαρμόζονται είναι η αναγκαιότητα για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων, το κατά πόσο δεν είναι υπερβολικά τα δεδομένα τα οποία ζητούν οι Αμερικανικές αρχές, να υπάρχει η αναλογικότητα. Όλες αυτές οι αρχές πρέπει να τηρούνται από τις χώρες μέλη. Συγχρόνως, οι εποπτικές αρχές είναι εθνικές. Δηλαδή την εποπτεία την κάνουν οι εποπτικές αρχές των χωρών μελών, οι εθνικές, η Ιρλανδική, η Γαλλική σε αυτή την περίπτωση και θα συμβούλευα τον αναφέροντα να έρθει σε επαφή με τις αρχές προστασίες δεδομένων, τις γαλλικές ή τις Ιρλανδικές ή και τις δύο και μπορεί να προσφύγει σε αυτές με καταγγελία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Λάνα Χέιρα. Καλησπέρα και από μένα. Από πλευράς φορολογίας τώρα. Αναφέρθηκε και πριν ότι η συμφωνία ΦΑΤΚΑ, οι συμφωνίε ΦΑΤΚΑ είναι διμερείς ανάμεσα στις ε, χώρες μέλη και τις ΗΠΑ. Δεν συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν παραβιάζεται λοιπόν το ευρωπαϊκό δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει να παίξει κάποιο ρόλο εδώ. Ανέφερε ο αναφέρον την εντολή για ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ελβετία, Μονακό, Σαν Μαρίνο κλπ. Είναι αλήθεια, αλλά για αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εντολή που τις είχε αναθέσει οι χώρες μέλη για να διαπραγματευτεί τέτοιες συμφωνίες. Το πεδίο εφαρμογή όσον αφορά τις πληροφορίες όμως θυμίζει πάρα πολύ τις συμφωνίες ΦΑΤΚΑ γιατί πρόκειται για διεθνή πρότυπα που βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στις συμφωνίες ΦΑΤΚΑ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στη συζήτηση. Οι συνάδελφοι τώρα. Η κυρία Ενχερβέλτ πρώτα απ' όλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να πω ότι ό,τι και να πω τώρα δεν είναι εναντίον των τριών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και συνειδητοποιώ ότι εσείς μεταφέρετε το μήνυμα. Οπότε δεν θα πυροβολήσω αυτό που φέρνει το μήνυμα. Αλλά όσα μας είπατε είναι μπουρδες. Απλώς και μόνο μπουρδες. Εγώ ε, πέντε χρόνια τώρα παρακολουθώ αυτή την υπόθεση. Και από το Μάρτιο του 2012 υποβάλλω προφορικές ερωτήσεις. Οπότε έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας λέει αυτά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Μας λέτε μετά δεν ξέρουμε, στείλτε μας πληροφορίες. Α, ναι, νομίζετε ότι τα δικαιώματά σας προστασία δεδομένων παραβιάζονται. Α, ενημερωθείτε και ειδοποιήστε τον εθνικό σας επόπτη. Όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως μας τη δίνει γιατί χρησιμοποιεί τις αρμοδιότητές της όποτε θέλει και τις υπερβαίνει επίσης όποτε θέλει. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί δεν υπάρχει νομική βάση για να πούμε στους Αμερικανούς όχι δεν μπορείτε να έχετε απρόσκοπτη πρόσβαση στα δεδομένα των Αμερικανών που ζουν στην Ευρώπη, αλλά ναι όταν πρόκειται για την Τουρκία. Δεν υπάρχει νομική βάση ούτε για το Fiscal Compact. Οπότε ειλικρινά κάνετε ό,τι θέλετε. Διαλέγετε και παίρνετε. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ είναι ότι κάθε φορά οι Ηνωμένε Πολιτείε χοροπηδάνε, η Επιτροπή τη λέει ναι βεβαίω. Μα οι διεθνεί σχέσει κάθε φορά παραβιάζουν τελικά τα δικαιώματα των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκτελεί τα χρέη τη. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί, να δούμε πώ λειτουργεί αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει να ονομάσει τον εαυτό τη Πολιτική Επιτροπή. Είσαστε όμω τόσο τεχνοκρακάτε που δεν είναι πιάστη. Και δεν το λέω για εσά, είπαμε, το λέω για τα αφεντικά σα. Εσεί θα πρέπει να στηρίζετε και να προστατεύετε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό πρέπει να κάνει η Επιτροπή. Εγώ δεν θέλω να ακούω τέτοια άλοθη χρησιμοποιείται νομικίστικα επιχειρήματα. Μπούρδε. Δεν ξέρω πόσοι τέτοιοι Αμερικανοί που έχουν γεννηθεί κατά λάθο στι Ηνωμένε Πολιτείε ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δικαιώματά του παραβιάζονται, μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό και όχι μόνο απλώ λογαριασμό. Γιατί να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε άλλα οικονομικά προϊόντα. Επειδή τυχαίνει να έχουν την Αμερικανή υπηκότητα γιατί εδώ δεν πρόκειται μόνο για την υπηκότητα. Δεν ξέρω, παιδιά που σπουδάζουν στις ΗΠΑ, τι έγκλημα έχουν κάνει. Γιατί πρέπει να αποκλείονται από άλλες υπηρεσίες. Εσείς το θεωρείτε φυσιολογικό. Μα μπορείτε να φανταστείτε εσείς να μην είχατε πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες. Τι θα σκεφτόσαστε για τα δικαιώματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν μπορούσατε να ζήσετε μια φυσιολογική ζωή γιατί τα θεωρείτε δεδομένα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αυτές οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι, μάλλον το πω είναι κάθε άλλο παρέκανοποιητικές. Επιμένω να πάμε σε ψηλότερο επίπεδο. Η αναφορά αυτή να μην κλείσει, να παραμείνει ανοιχτή, να παρακολουθήσουμε σε πολιτικό επίπεδο την εξέλιξη και να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει από το σπίτι αυτό να ξεκουμποθεί και να φροντίσει να βρει μια καλή λύση για αυτή την υπόθεση που τραβάει εδώ και χρόνια. Δεν είναι από το Σεπτέμβριο, είναι για χρόνια που αποκλείονται οι άνθρωποι αυτοί από βασικές οικονομικές υπηρεσίες. Και αυτό είναι το χρέος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν είναι απρόθυμη να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών της Επιτροπή, ε, να πάει σπίτι της και για να είμαι ειλικρινή, αν δω πώ κάνει η πολιτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλο και περισσότερο έχω όρεξη να προτείνω να πάνε σπίτια του. Γιατί αρνούνται να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά του. Εγώ έτσι αισθάνομαι, κυρία Πρόεδρε, και ήθελα να το έχω πει. Ευχαριστούμε πολύ όλοι μου φαίνονται προβληματισμένοι και νομίζω έχουν πάθει σοκ. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να το χωνέψουμε όλα αυτά. Θέλετε να εξηγήσω, λέει η κυρία Νετβέλτ. Όχι, όχι, λέει η πρόεδρο, όχι αυτή τη στιγμή. Το μήνυμά σα ήταν σαφέστατο, πρέπει να πω. Θα ήθελε κάποιο άλλο να πάρει το λόγο. Όχι. Ούτε εσεί, για Τι γίνεται εδώ. Ωραία λοιπόν, να σε επιστρέψουμε στον αναφέροντα. Έχετε το λόγο για άλλα δύο λεπτά. Υπογραμμίστε τι θέλετε να κάνουμε. Η Σοφή το είπε πολύ καλά. Για να σας το δώσω ε, ε, πιο παραστατικά. Έχουμε χιλιάδε τέτοιου κατατύχει Αμερικανού. Και αυτό που είναι τρομακτικό με το ΦΑΤΙΑ και δεν καταλαβαίνει η Κομισιόν δεν είναι μόνο οι κατατύχοι Αμερικανοί, των οποίων οι πληροφορίε δίνονται στην Αμερική. Ένα Γερμανό τυχαίο Αμερικανό ε, έχει την κυδαιμονία των λογαριασμών τη μητέρα του, η οποία πεθαίνει και το γεγονός ότι ελέγχει αυτούς τους λογαριασμούς της γερμανίδας μητέρα του, σημαίνει ότι αυτή η Γερμανίδα 20 που δεν έχει καμία σχέση με την Αμερική, ε, ε τα στοιχεία της πάνε στο IRS. Αυτό δεν είναι παραβίαση του άρθρου 8. Και έχουμε χιλιάδες τέτοια παραδείγματα. Οπότε επαναλαμβάνω το αίτημά μου. Θέλουμε η Κομισιόν να ζητήσει εντολή, όπως έκανε με την Ελβετία και το Μονακό, να αναθεωρήσει το ΦΑΤΚΑ για εκ μέρους όλων των κρατών μελών με τις Ηνωμένε Πολιτείες ώστε να υπάρξει αμοιβαιότητα, να εφαρμοστεί η αμοιβαιότητα αυτή ε, ε, και επειδή δεν εφαρμόζεται μπορούμε να επανέλθουμε σε διαπραγματεύσεις. Αυτό πρέπει να γίνει και αυτό χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας, ε, όχι μόνο εσάς αλλά και τους ε, φίλους κατά τύχη Αμερικανού σα και ευχαριστούμε που επισημάνετε τη σπουδαιότητα αυτού του θέματο. Έχει έρθει η ώρα να το συνοψίσουμε. Δεν είναι εύκολο. Η κυρία Νετφέλτ έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να το στείλουμε σε υψηλότερο επίπεδο, πολιτικό επίπεδο και μπορούμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμεί ε, ω Επιτροπή Αναφορών είναι να αφήσουμε φυσικά ανοιχτή την αναφορά και εγώ θα την επαναφέρω στους συντονιστές για να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη τις νομοδοτήσεις της ΕΚΟΝ και της ΛΥΜΠΕ είναι αρκετά ε, ε, σαφές το μήνυμα εκεί και να ξεκινήσουμε μια συζήτηση στην Ολομέλεια βάσει αυτών. Δεν μπορώ να σα το υποσχεθώ αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό μπορώ να κάνω να το ξανασυζητήσουμε με τους συντονιστέ, να υπογραμμίσουμε το πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Συμφωνείτε? Ωραία. Αφού γνέφουν όλοι από όλε τι ομάδε, είμαι ασφαλή. Οπότε ούτω και θα πράξουμε και προχωράμε παρακάτω. Περνάμε λοιπόν στην ετήσια έκθεση, σχετικά με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητού. Η κυρία Μίτση είναι η συγγήτρια, έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου δίνετε το λόγο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτή την ε, έκθεση, όπως ε, είπα, ε, και όταν ήταν εδώ μαζί μας η διαμεσολαβήτρια η κυρία Αράλη εγκρίνουμε στη δική μας έκθεση τα όσα έχει κάνει η διαμεσολαβήτρια είναι καλά συνταγμένη η συγκεκριμένη έκθεση δεν πρόκειται δηλαδή για μια έκθεση την οποία κάποιο συνδυάζει και την οποία δεν αντιλαμβάνεται κανεί. Έχει κάνει πραγματικά εξαιρετικό έργο εδώ η κυρία Οράιλη. Ε, δεν θα συνοψίσω ε, τα όσα περιλαμβάνει αυτή η έκθεση. Απλώ θα σα αναφέρω τα όσα εγώ προτίθεμαι να συμπαραλάβω στη δική μου έκθεση σε ό,τι αφορά την έκθεση τη Διαμεσολαβήτρια. Οι κύριε λοιπόν συστάσει που κάνω ε, στη δική μου έκθεση είναι να συνεχίσουν οι στρατηγικές έρευνες σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια της Επιτροπής, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ε, των ε, καταγγελιών για διαδικασία κατά παράβαση το 2017, να συνεχίσουν οι ε, διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά τους τριμερείς διαλόγους και οι διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του Βασίλειου, να συνεχίσει τη εργασία σε ό,τι αφορά την ε, διαφάνεια τη οικονομική ολοκλήρωση και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα στο πλαίσιο τη ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ε, τη ECT, και να συνεχίσει τη συνεργασία τη και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμακευτικών Προϊόντων, προκειμένου να συνεχίσει η διασφάλιση τη υψηλή ποιότητα των δοκιμών στι οποίε προβαίνει. Επίση, υπάρχουν και κάποιε συστάσει προ την Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα, με βάση ακριβώ τα όσα αναφέρει η έκθεση τη διαμεσολαβήτρια. Αναφέρουμε δηλαδή ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν οι συστάσει ε, ε, τη διαμεσολαβήτρια ε, και ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί δηλαδή η Επιτροπή στι υποχρεώσει τη, όπω βγάζουν από τι συνθήκε. Εδώ αναφέρομαι ειδικότερα Ε, στην ε, ανάληψη επαγγελματικών ε, καθηκόντων, δηλαδή θέσεων εργασία από την πλευρά των επιτρόπων, με μετά την άλλη, ενώ υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Επίση, καλείται η Επιτροπή να εφαρμόσει τι συστάσει τη διαμεσολαβήτρια σε ό,τι αφορά ε, τον ε, διορισμό των ε, ειδικών της και τον, τον διορισμό των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Αυτές λοιπόν είναι οι συστάσεις Διαμεσολαβήτρια, τις οποίες υποστηρίζουμε, αλλά από εκεί και μετά αναμένουμε ενδιαφέρον και τη συνέχεια που θα δώσει, στις δράσεις δηλαδή στις οποίες θα προβεί η διαμεσολαβήτρια, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το πώς οι κανόνες που ισχύουν σήμερα, τα soft rules, ρυθμίζουν ακριβώς αυτήν την ανάληψη ε, των ε, πολιτικά εθνότων από την Επιτροπή ε, Αντίστοιχων Επαγγελματικών Θέσεων. Και επίσης ε, η ε, εφαρμογή των, ε, και η συμμόρφωση με την, Ευρωπαϊκή, με την Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι κάτι που μα ενδιαφέρει με βάση και τα όσα έχει προτείνει και η Γενική Διεύθυνση ΣΑΚΟ σε σχέση με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των κανονικών προϊόντων. θα μπορούσαν δηλαδή να εφαρμοστούν όλα τα σημεία της Ανόγου από τη δική μας πλευρά. άρα λοιπόν η δική μα έκθεση θα ανακεφαλαιώνει τι προηγούμενε συστάσει που έκανε διαμεσολαβήτρια σε ό,τι αφορά ειδικότερα την περαιτέρω συζήτηση της Ευρωπαϊκής, για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, την οποία θα συζητήσουμε και εδώ στη συνέχεια. Και επίση αναφέρουμε ε, τα όσα ε, αναφέρονται σε σχέση με του πληροφοριοδότε ε, με, με, που παρέχουν πληροφορίες μεγάλης ε, πολιτικής ε, σημασίας, δηλαδή το πώς ε, μπορεί περαιτέρω να αυξηθεί η προστασία των λόγων προσώπων, όπως είναι γνωστά ως whistleblowers. Άρα λοιπόν, οποιασδήποτε τροποποιήσεις τώρα γίνουν, θα γίνουν ενδεχομένως μέσω τροπολογιών. Τώρα, ημερομηνίε. Στις 11 Ιουλίου θα γίνει συζήτηση στην ειδική μας Επιτροπή Αναφορών. 18 Ιουλίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στις 3 το μεσημέρι και 11 με 12 Οκτωβρίου κανένα λάθος είναι ψηφοφορία στην δική μας ε, Επιτροπή για το αναφορών και συνέχεια βέβαια ψήφιση στην Ολομέλεια. Ευχαριστούμε Λένα Πολύ καθαρή επισκόψη του περιεχομένου της έκθεσης. Ο Γέρακ έχει ζητήσει τον λόγο ο Σκιώδης ε, εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Ναι, σωστά είπατε κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Εκ μέρους της ομάδας του ΕΛΚΑ ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Συγήτρια για την εκπόνηση αυτής της ε, πλήρους ε, περιεκτικής έκθεσης. Είναι ισορροπημένη, καλαδομημένη και περιγράφει ό,τι είναι σημαντικό για το έργο του Ευρω... της Ευρωπαϊκής Λαβήτριας και του γραφείου της. Εγώ παρακολουθώ το έργο της κυρίας Ωραίλη από την αρχή και πρέπει να πω ότι οι ιδέες της έχουν συμβάλει στο να γίνει αυτό το γραφείο πιο φιλικό προς τους πολίτες και πιο ευκολονόητο. Η προσέγγιση αυτή είναι ορατή σε όλο το υλικό που δημοσιεύεται από τότε που ανέλαβε καθήκοντα η κυρία Ωραίλη. Αλλά και στη στρατηγική επικοινωνία ε, είναι αυτό ορατό και σε εκδηλώσει που διοργανώνονται Πιστεύω ότι στις δύσκολες εποχές που ζούμε σήμερα είναι ύψης της σημασίας ε, να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών. Είμαι της άποψης ότι το γραφείο αυτό συμβάλλει ακριβώς σε αυτό. Και αυτό εκφράζεται με ρυθμούς. Ε, ο αλληλεπιδραστικός οδηγός, χάρη στον οποίο όλοι μπορούν να πλογηθούν μόνοι της για να βρουν το όργανο που χρειάζονται, αξίζει συγχαρητήρια. Ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που ανέφερε τι διαδικασίε επαναβάσεις στο σημείο 8. Κατά την άποψή μου είναι πράγματι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τις προσπάθειες της Κομισιόν να διευκολύνει την πρόσβαση στα έγγραφα και τις πληροφορίες ειδικότερα όσον αφορά διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με αναφορές που έχουν ληφθεί Ενθαρρύνει επίσης ε, τη συνέχιση των στρατηγικών ερευνών της Δημοσιολαβήτριας για θέματα διαφάνειας της Κομισιόν ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση των ε, παραπώνων για περιπτώσει παράβασης. Εγώ προτείνω να παρακολουθούμε τακτικά το ζήτημα αυτό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο σημείο 9 που αφορά τη διαφάνεια στις εμπορικές συμφωνίες και διαπραγματεύσεις. Η διαφάνεια και επικοινωνία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ζωτική σημασία για τους πολίτες μας, ειδικότερα ε, αν παρατηρήσει κανείς ε, τι έχει συζητηθεί κατά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις τέτοιου είδους. Ωστόσο αυτή η διαφάνεια δεν πρέπει να υπονομεύει τη διαπραγματευτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε μια σωστή ισορροπία. Θέλουμε διαφάνεια μεν, αλλά όχι αυτή η διαφάνεια να υπερβαίνει κάποια όρια και να υποβαθμίζει τη διαπραγματευτική μας θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μπέτρις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκ μέρους του Χαβιέρ Νατ, που είναι ο Σκιώδης για την Άλντε, θέλω να ευχαριστήσω τόσο την εισηγήτρια, όσο και τη συνηγόρα του πολίτη για την άλλη. Οι τροπολογίες μας θα μιλήσουν για περισσότερη διαφάνεια και στο Συμβούλιο Υπουργών στις διάφορες συνεδριάσεις, όλα και στα πρακτικά. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ποιοι βρίσκονται τριγύρω. Η πρόσβαση σε έγγραφα επίσης πρέπει να είναι άμεση και χωρίς καθυστερήσεις που φτάνουν 6 μήνες μερικές φορές θεωρούμε ότι είναι βασικό η ετήσια συνεδρίαση των ε, συνηγόρων του πολίτη να γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Επιτροπή δεν έχει να προσθέσει τίποτα, οπότε δίνω το λόγο και πάλι σε σένα, Μαρλένα, αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Προσβλέπω σε καλή συνεργασία με τους σκιώδεις. Καλώς να ξέρετε ότι μέχρι τις 18 Ιουλίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 3. Η συνήθις διαδικασία. Και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η γνωμοδότηση για την αναθεώρηση του κανονισμού 211 του 2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών. Η συγητής είναι ο κύριος Βαλέσα. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό που συζητούμε την αναθεώρηση αυτή της πρωτοβουλίας πολιτών εδώ στην Επιτροπή μας. Η ΑΦΚΟ, η Επιτροπή Σταματικών Υποθέσεων, είναι επί της ουσίας αρμόδια και υπάρχει και κάτι που και αυτή παρεμβαίνει. Εμείς λειτουργούμε βάσει ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος προκειμένου να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χρησιμοποιήσει καλύτερα αυτό το τόσο χρήσιμο εργαλείο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι τα τέλη της εβδομάδας αυτής και μόνο στα αγγλικά. Ξέρω ότι δεν είναι η καλή, σωστή διαδικασία, αλλά δεν έχουμε χρόνο για να το κάνουμε αλλιώς. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδες εισηγητές για την καλή συνεργασία που είχαμε. Η εβδομάδα 36η φαίνεται ότι είναι η καλύτερη για να προβλέψουμε συνάντηση των σχεδόν εισηγητών και η γραμματεία θα είναι σε επαφή μαζί σας με μια συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα για την γνωμοδότηση έχουμε ελάχιστα περιθώρια για να βάλουμε μέσα τα πάντα. Αλλά προτείνω 7, ε, σημεία. Πρώτον, το παραδεκτό. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια της διαδικασίας της λήψης αποφάσεων και να διευκρινιστεί ποια είναι τα κριτήρια για το παραδεκτό μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Δεν είναι πάντα ξεκάθαρο στις διάφορες ε, αποφάσεις. Πρέπει αυτές να καταγράφονται. Η Επιτροπή πρέπει να κωδικοποιήσει επίσης τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με πρωτοβουλίες μειονοτήτων. Δεύτερον, η διαδικασία. Πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ευκολή φιλική προς το χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς και νομικούς περιορισμούς και να απλοποιείται η όλη διαδικασία με την ηλεκτρονική υπογραφή. Να μην υπάρχουν πια τα τεχνικά προβλήματα και δυσκολίες για να λαμβάνεται υπόψη η συλλογή αυτή των υπογραφών και ηλεκτρονικά. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να δει τις διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τα δεδομένα στα διάφορα εθνικά συστήματα. Η υπηκότητα, για παράδειγμα, ε, τόπος διαμονής προτείνω, μάλλον συμφωνώ και εγώ με την πρόταση της ΑΦΚΟ που αναφέρεται σε ένα κεντρικό σύστημα συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών. Να χρησιμοποιεί προτείνω τις τεχνολογίες τις ήδη υπάρχουσες για πλατφόρμες έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η συλλογή ηλεκτρονικών πληροφοριών. Και είναι ζωτική σημασία να υπάρχει και περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τα χρηματοδοτικά, τη χρηματοδοτεί την κάθε τέτοια πρωτοβουλία. Τρίτον, one stop shop. Όντως, θα πρέπει να υπάρχει ένας μόνος τρόπος να προχωρήσει κανείς βήμα το βήμα. Να υπάρχει μία θηρίδα εντό εισαγωγικών ε, από την οποία μπορεί να ενημερωθεί ο πολίτης για την πρωτοβουλία. και να υπάρχει νομική βάση για περίπτωση καταγγελιών. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει αυτή η νέα θηρίδα. Τέταρτον, να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό. Στηρίζω και άλλη μια φορά την πρόταση της ΑΦΚΟ, ώστε να παρακολουθούμε τι γίνεται τελικά με αυτές τις πρωτοβουλίες πολιτών που έχουν προχωρήσει, που είναι επιτυχείς. και να φροντίσει γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης. Με στην πρώτη γραμμή τις επιτροπές που είναι αρμόδιες για τα θέματα για τα οποία είναι αυτές οι πρωτοβουλίες, συν τη δικιά μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Κατά τη γνώμη μου, οι δημόσιες ακροάσεις θα πρέπει να επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, των εμπειρογνωμόνων, των ε, όσων έχουν συμμετάσχει στην πρωτοβουλία. Και να αποζημιώνονται τα έξοδα ταξιδιών τους όπως κάνουμε και με τους αναφέροντες. Και πέμπτον, λόμπις. Εδώ θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα που θα έπρεπε να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων από τη μία πρέπει να αποφασίζουν για το παραδεκτό ή όχι και μετά πρέπει να φροντίζουν και για την διοικητική συνέχεια και τη διεξαγωγή. Δεν μπορεί να τα έχει όλα αυτά στα χέρια της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων εδώ. Τέλος, ζητώ συγγνώμη που το χρονοδιάγραμμα είναι τόσο σφιχτό, αλλά προσβλέπω πάντως τη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε το λόγο στους συναδέλφους. Κυρία Μπεσαρέκτη, το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Ο εισηγητής ο κύριος Βαλέσα νομίζω ότι πολύ καλά παρουσίασε τα διάφορα θέματα που μας απασχολούν. είναι αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη έκθεση που κάναμε την ΑΦΚΟ για την αναθεώρηση της πρωτοβουλίας πολιτών. Απλώς προσθέτω την ανησυχία της Άλντε για το θέμα ακριβώς του παραδεκτού και επίσης και κυρίως για την αποτελεσματικότητα. Πρέπει να απαντάμε με το χέρι στην καρδιά στους πολίτες η προσοχή μας να είναι πλήρης και να είμαστε αποτελεσματικοί, εξού και η ενία θηρίδα, που μπορεί να εφαρμοστεί πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας εγκαταστάσεις που διαθέτουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε όλες τις πρωτεύουσε. Οπότε εύκολα μπορεί να το πείσει κανείς που βρίσκεται αυτή η ενία θηρίδα. Είναι μια σημαντική στιγμή για να ευθυγραμμίσουμε την απάντησή μας όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και να δώσουμε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την αναθεώρηση αυτής της πρωτοβουλίας που ήταν μια από τις πιο σαφείς υποσχέσεις που κάναμε στους πολίτες. Το λέμε και στην έκθεση για την Ευρωπαϊκή Θαγένεια που ετοιμάζουμε. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε αυτό που ονομάστηκε αδιαφυσβήτητο εργαλείο υπέρ των πολιτών να καταλήξει σε μια αποτυχία. Ευχαριστούμε η κυρία Μίτσα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαλέσα για αυτή την έκθεση είναι πολύ πλήρης γνωμοδότηση, ε, είναι περίπλοκο το θέμα. Ε, με το οποίο δεν ήταν εύκολη να ασχολήσει. Τα κατάφερα όμω πολύ καλά και πολύ ισορροπημένα ο κ. Βαλέσσα. Ενισχύει και τη θέση της Πέτη που είχαμε πριν από δύο χρόνια. Υποστηρίζω την προσέγγιση του κ. Σιγητή. Ε, χρειάζεται πράγματι μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων μεγαλύτερη απλούστευση της ε, online συλλογής υπεγραφών και της ε, προοδευτικής προσέγγισης άρσης των τεχνολογικών εμποδίων αλλά και το One Stop Shop για ECI και η πρόταση ε, παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των ECI. Αυτό είναι πολύ καλό των πρωτοβουλίων. Έχω μια παρατήρηση. Δεν είμαι βέβαιος αν γίνεται για τις προτάσεις ΑΦΚΟ. Αναφέρεστε στην τωρινή έκθεση ΑΦΚΟ. Δεν μπορούμε να κάνουμε αναφορά σε κάτι το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή και δεν έχει ακόμα ψηφιστεί. Εγώ λοιπόν θα υποβάλω κάποιες ε, τροπολογίες γι' αυτό, διότι πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίζουμε ότι αυτή τη φορά η Επιτροπή θα θα απλουστεύσει πράγματι τι πρωτοβουλίες χωρίς να επιστρέφουμε ξανά μετά από δύο χρόνια για να απλουστεύσουμε πάλι τα πράγματα. Ε, χρειάζεται μια πιο διαφανής διαδικασία για την καταχώρηση και χρειαζόμαστε σαφή καθορισμό του πεδίου ε, εφαρμογής των ε, πρωτοβουλίων. Χρειάζεται πιο συνεκτική προσέγγιση, ε, ειδικότερα όταν δίνεται αιτιολόγηση απόρριψης κάποια πρωτοβουλία. Ε, χρειαζόμαστε και περισσότερη προβολή των πρωτοβουλειών ε, στο κοινό, στα μέσα διότι έχω την αίσθηση ότι οι πολίτε δεν γνωρίζουν αρκετά για τι πρωτοβουλίε των πολιτών. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυτού να τι αξιοποιήσουν. Υπάρχουν και κάποια τεχνικά ζητήματα, απαιτήσει στοιχείων, ε, ηλεκτρονικέ διαδικασίε, ε, η 12μηνη περίοδο συλλογή υπογραφών. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εκεί θα επικεντρωθώ εγώ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστούμε πολύ καλά. Ο κ. Τερικάπρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιγητή για την εξαιρετική του γνωμοδότηση. Εγώ πιστεύω ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες ε, στο σχεδιασμό των πρωτοβουλίων των πολιτών είναι τρεις. Περιοριστική διαδικασία καταχώρησης, δεύτερον ε, έλλειψη παρακολούθηση από την Κομισιόν και τρίτον δύσκολη διαδικασία συλλογής υπογραφών. Ο εισηγητής ε, ε, έχει ασχοληθεί με το τελευταίο πρόβλημα πολύ σωστά. Εγώ θα υποβάλω κάποιε τροπολογίες που αφορούν τις σημερινέ. ελλείψεις και να αναφέρω τώρα κάποιες από τις τροπολογίες μου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπάρχει ένας ανεξάρτητος φορέας που θα πραγματοποιεί τον αρχικό έλεγχο για την καταχώρηση αποφεύγοντας έτσι τις συγκρούσεις συμφερόντων της Κομισιόν. Δεύτερον, θα ήθελα να επιτρέπονται πρωτοβουλίες ε, που να απαιτούν αλλαγές στις συνθήκες που πλέον δεν είναι ούτε αδύνατες ούτε παράνομες. Τρίτον, θα διευκόλυνα τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οποιασδήποτε από τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών. Τέταρτον, θα αύξανα τη διαφάνεια και την ποιότητα των ελέγχων χρηματοδότησης και χορηγίας των πρωτοβουλίων. Και πέμπτον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για εσάς, το ξέρω ότι μας το είπατε, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό σημείο, θα διασφάλιζα ότι η Κομισιόν θα έκανε μια νομοθετική πρόταση, εγώ θα έλεγα εντός μετά από την υποβολή μιας επιτυχούς πρωτοβουλίας. Για την παρακολούθηση, διότι αν δεν γίνει τίποτα και απλά ο κόσμος μαζεύει υπογραφές ε, ε, και κάνει τόσο κόπο για όλα αυτά, για να συλλέξει υπογραφές ε, ανά την Ευρώπη και μετά η Κομισιόν απλά συλλέγει υπογραφές. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, ούτε είναι πολύ καλό αυτό για τους πολίτες μας. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που είχε πει ο Τίμερμαν μια φορά εδώ στο κοινοβούλιο πριν από λίγες εβδομάδε. Είπε μην έχετε και υπερβολικέ προσδοκίε για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Αυτό δεν μας καθησυχάζει, ούτε μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα. Γι' αυτό το λόγο εύχομαι σε εσά κύριε Βαλέσα και εύχομαι για όλους μας και σε όλη την ομάδα. Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, συμπεριλαμβάνεστε και εσείς αυτό, ε. Ας πάμε στον εισηγητή, αν έχετε να πείτε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το εργαλείο. Το καταλαβαίνουμε όλοι εδώ και για να το βελτιώσουμε έχουμε διάφορες θέσεις, αλλά γενικά όλοι συμφωνούμε ότι κάποια πράγματα μετά από δύο χρόνια μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν. Χαίρομαι λοιπόν που μπορούμε να βρούμε ε, κοινό τόπο στο περισσότερα θέματα. Ε, το ανεξάρτητο οργανισμό τώρα, το ανεξάρτητο φορέα, δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσει ποτέ η Κομισιόν με αυτό, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε. Γιατί ναι, προφανώ υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, αλλά ναι, εγώ προσβλέπω στι ε, τροπολογίε σα και είμαι βέβαιο ότι θα μπορέσω να συμφωνήσω μαζί σα στι περισσότερε. Ευχαριστώ. Πολύ καλά, Πρόεδρος. Και τώρα πρέπει να σας πω ότι η προθεσμία τροπολογιών είναι Παρασκευή 14 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι. Στα αγγλικά μόνο όπως ζήτησε ο εισηγητής και πολύ σημαντικό η 84 EM δεν θα είναι διαθέσιμη. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω εγώ. Οι 84 τροπολογίες δεν θα είναι διαθέσιμες, θα πρέπει να τις δώσετε ε, μη αυτόματα. Ε, καλό είναι να ξέρει κανείς πώς θα το κάνει αυτό. Και εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή συνάντηση. Το πιστεύετε ή όχι, η επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα 7 Σεπτεμβρίου, ολοήμερη. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, φάτε πολύ παγωτό, κολυμπήστε πολύ στη θάλασσα και ελάτε ακόμη πιο όμορφοι από ό,τι είστε σήμερα.